warm welcome, uh, dear colleagues. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, ευρωβουλευτές, αγαπητά μέλη από τις Εθνικές Βουλές, ε, κύριε Επίτροπε, αγαπητέ κύριε Τσβετάνοφ, ε, κυρία Σαχίν, ε, δήμαρχε, κύριε και εισηγητά των Ηνωμένων Εθνών Κοσάλες, κύριε Υπουργέ Βέμπερ, Καλωσορίζουμε φυσικά και την ε, Βουλγαρική Προεδρία στη συνεδρίαση και θερμό καλωσόρισμα σε όλους τους εξέχοντες ε, καλεσμένους μας. Εγκάρδια σας καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Εμείς στην Πολιτική Πολιτικών Ελευθεριών, όπως γνωρίζετε, πραγματευόμαστε μερικά από τα πιο δύσκολα και ευαίσθητα ζήτηματα ε, της εποχής μας και η μετανάστευση είναι ένα από αυτά και στη διακοινοβουλευτική αυτή σύσκεψη για το θέμα της μετανάστευσης ε, τους ε, νόμους διάβλους και την ένταξη θέλουμε να έχουμε μια καρποφόρα ανταλλαγή απόψε μεταξύ μας και σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είναι μαζί μας σήμερα 39 μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων από 16 διαφορετικά κράτη-μέλη και μάλιστα και από την Ορβηγία, μια χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Κάτι που είναι περίτρανη απόδειξη του ζωηρού ενδιαφέροντο που προκαλεί το σημερινό θέμα. Επίση, ε, έχουμε και δύο ομάδε καλεσμένων από την Κάμπια και την Τουρκία. Και φαντάζομαι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εθνικών βουλευτών και των ευρωβουλευτών για του ε, νόμιμου διάβλου και την ένταξη των μεταναστών σχέση με το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση είναι ένα πολύ επίκαιρο και πολύ ευαίσθητο θέμα. Και μάλιστα τα δύο ζητήματα φαίνεται ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας και πολιτικής συζήτησης στα κράτη-μέλη. Εμείς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ασχολούμαστε ιδιαίτερα με τα θέματα αυτά, αλλά δεν θα έχει κανένα νόημα χωρίς βαθιά κατά ε, συνεννόηση και συζήτηση με τα κράτη-μέλη. Και σήμερα στην διακοινοβουλευτική αυτή σύσκεψη θα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να συζητήσουμε ευρωβουλευτές και εθνικοί βουλευτές εκτενέστατα μαζί με εκπροσώπους θεσμικών οργάνων, φορέων, οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, πανεπιστημιακών, εμπειρογνωμών και το καθεξής. Και από κοινού θα κάνουμε ένα απολογισμό της απάντησης στις προκλήσεις της μετανάστευσης, όπως αναφέρεται αρχικά στο κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το θεματολόγιο και τη μετανάστευση του 2015. Και χαίρομαι ιδιαίτερω που είναι μαζί μα σήμερα ο Επίτροπο Αβραμόπουλος. Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό εδράζεται στα στου τέσσερι πυλώνε για την καλύτερη διαχείριση τη μετανάστευση. Στο θεματολόγιο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση με προτάσει για την αντιμετώπιση τη παράτυπη μετανάστευση, ενίσχυση τη κοινή διαχείριση των συνόρων, τη ενίσχυση τη κοινή πολιτική ασύλου και της, ε, των, ε, της ε, θέσπισης νέας πολιτικής για τη μετανάστευση. Ε, αυτά είναι στη θεωρία. Στην πράξη όμως τι πετύχαμε. Αυτό θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευρά του, εδώ στην Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών, επίση διατράνωσε τη θέση του στο ψήφισμα του Απριλίου του 2016 για την κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη μια σφαιρική ε, πολιτική ε, μεταναστευτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να μην ξεχνούμε και τι μακροπρόθεσμε προοπτικέ τη μετανάστευση και κυρίω τι ανάγκε τη μεταναστευτικέ δεδομένη τη γύρανση του πληθυσμού και της οικονομικής δραστηριότητας. Και μάλιστα αυτά θα πρέπει να παρεμποδίζει την ανάγκη της δημιουργίας νόμιμων διάβλων ε, μετανάστευσης και της διευκόλυνσης ε, της, πολύ σημαντικής ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία για να διαχειριστούμε καλύτερα την κινητικότητα και μάλιστα με πιο βιώσιμο και αηφόρο τρόπο. Το ψήφισμα επίσης ε, λειτουργεί ως πηξίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στις διαπραγματεύσεις για τη μεταρρύθμιση του κοινού συστήματος ασύλου. Και αυτό το θέμα μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα σήμερα. Η πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος της μπλε κάρτας. Είναι κάτι που, όπως ξέρετε, έτυχε ένθερμης υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποτελεί ένα παράδειγμα του πού εντοπίζονται τα σοβαρά προβλήματα στα κράτη-μέλη. Και αυτό είναι κάτι που έχει και συμβολική αξία ε, και είναι δεικτικό του, ε, της πρόοδου που πραγματοποιούμε ή όχι στα θέματα των διάβλων. Οπότε τα ερωτήματα είναι... Το Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για τη Μετανάστευση έχει αποφέρει αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις νόμιμες διόδους και την καλύτερη ένταξη των μεταναστών. Τι έγινε με τις λεγόμενες ε, νόμιμες διόδους ή τους νόμους διάβλους ε, μετανάστευσης. Πού έγκυται η νέα πολιτική για την, παράνομη, για την νόμιμη συγγνώμη, μετανάστευση. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υιοθετεί μέτρα και στηρίζει καλύτερα την ένταξη των προσφύγων στα κράτη-μέλη. Αυτά τα ερωτήματα καλούμαστε να απαντήσουμε σήμερα και θα ήθελα να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Τσβετάνοφ, τον πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικών Υποθέσεων και Δημόσιας Τάξης της Βουλγαρικής Βουλής και με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να του δώσω το λόγο για, μια... για την ομιλία του. Κύριε Σβετάνοφ, σας ευχαριστώ που ήρθατε και έχετε το λόγο. Αγαπητέ κύριε Αβραμόπουλε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, αξιότιμα μέλη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τις προσπάθειές σας. Προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να επανέλθει η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της μετανάστευσης σε ε, φυσιολογικά επίπεδα. Θα θυμάστε τι είχε συμβεί μετά το 2011 και την Αραβική Άνοιξη και στη συνέχεια μετά τον πόλεμο της Συρίας. Το 2015 τις μεγάλες μεταναστευτικές ροές που ακολούθησαν. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας ε, εξηγήσω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι αφού υιοθετήθηκε το Μάιο του 2015 η Συμφωνία για τη Μεταναστευτική Πολιτική, μπορέσαμε και μπορούμε σήμερα, δύο χρόνια μετά, να συζητούμε ε, πανευρωπαϊκά μέτρα ε, για να αντιμετωπιστεί ε, το πρόβλημα της μετανάστευσης και θέλω να υπογραμμίσω, στα όσα είπε και ο κύριος Μωράες, ότι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθούν νόμιμοι δρόμοι, νόμιμοι διάβλοι μετανάστευσης. Πρέπει να δοθούν λύσεις στα προβλήματα και ταυτόχρονα πρέπει να περιοριστεί και η παράτυπη μετανάστευση. Θα θυμάστε τι αντιμετώπισαν οι χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και άλλες χώρες μέλη οι οποίες ε, σήκωσαν μεγάλο βάρος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας εξηγήσω τι κάναμε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με την ε, Τουρκία, η οποία γνωρίζετε πως συμβάλλει στον περιορισμό των ε, ροών παράνομης μετανάστευσης. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία από πλευρά τους βεβαίως καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιμένουμε βέβαια να προχωρήσει το έργο σε άλλα νομοθετικά κείμενα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω αυτό που και ο κύριος Μωράες σε σχέση με την ε, υπόθεση, με την πρόταση για την μπλε κάρτα. Μαζί με άλλες προτάσεις θα μας επιτρέψει η πρόταση αυτή να προσελκύσουμε εργαζομένους με υψηλές δεξιότητες στην Ευρώπη, ανθρώπους οι οποίοι θα φέρουν προστιθέμενη αξία και βέβαια θα δώσουμε έτσι αποτελεσματική απάντηση και στους ε, λαϊκιστικούς ε, τόνους που διαδίδονται αυτή τη στιγμή, γιατί βέβαια ο λαϊκισμός τρέφεται από τις ροές της παράνομης μετανάστευσης. Ε, θέλω επίσης να συγχαρώ τον Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο για την προσήλωσή του, για τη βοήθειά του σε αυτή την, στο σχεδιασμό της μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι πολύ σημαντικός ε, ο ρόλος του. Τα εθνικά μας κοινοβούλια γνωρίζουν ήδη πως είναι ο κύριος Αβραμόπουλος ε, διατεθειμένος ότι ε, δέχεται οποιαδήποτε πρόσκληση για να πάει στα Εθνικά Κοινοβούλια να συζητήσει μαζί τους ποια είναι η καταλληλότερη πολιτική για τη δημιουργία των, ε, για την εξασφάλιση των νόμιμων εκείνων διάβλων που θα φέρουν ε, την ειρήνη και την ευημερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να ε, εστιάσουμε την προσοχή μας και στις συμφωνίες επανεισδοχής βεβαίως, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να περιορίσουμε τις ε, ε, ανεπιθύμητες μεταναστευτικές ροές, δηλαδή εκείνες τις οποίες οργανώνουν οι λάθροδιακινητές, αυτοί δηλαδή οι οποίοι κερδίζουν τεράστια ποσά από τη διακίνηση. Τι άλλο να προσθέσω εδώ. Κάποια λόγια ίσως για το κοινοβούλιο σας, επιτρέψτε μου. Ελπίζω ότι από κοινού με τον κύριο Μωράης και με όλους σας βέβαια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάθε πτυχή για τη μετανάστευση στη Σόφια σε ένα περίπου μήνα. Είμαι πεπισμένος πως από κοινού είμαστε πιο ισχυροί, μαζί είμαστε πιο ισχυροί. Ευχαριστώ τον κύριο Μωράης που εξασφαλίζει την το απαραίτητο κλίμα και τις συνθήκες εκείνες ε, πάντα συμβάλλει στην ε, οργάνωση έτσι ώστε να προχωρούμε όλοι ενωμένοι η μετανάστευση και όλα όσα πράττουμε για να, την, για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη μετανάστευση, ξέρετε ότι θα είναι ένα από τα κύρια ζητήματα που θα μας ε, συνοδεύσουν έως τις επόμενες ευρωεκλογές, έως το 2019. Και κύριε Πρόεδρε, αυτά είχα να πω Σταματώ εδώ. Και ελπίζω όλα τα κοινοβούλια να συμβάλλουν και να συνεχίσουν να συμβάλλουν στις συζητήσεις για το θέμα της μετανάστευσης αλλά και σε όλα τα συναφή ζητήματα, οδηγία για την μπλε κάρτα και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε όλα τα ζητήματα να αντιμετωπιστούν και πάνω απ' όλα να ενσωματωθούν στις κοινωνίες μας όλοι οι αλλοδαποί που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Να αναφέρω ότι ε, λαμβάνει χώρα πριν από το Συμβούλιο ε, και Θαλαβόγαρ στη Βουλγαρία, όπου θα συζητηθούν αυτά τα θέματα. Ξεκινάμε λοιπόν με την πρώτη, την πρώτη φάση που θα εστιάσει στις, ε, στους νομικές διάβολους και στην ένταξη. Είναι τιμή μου να καλωσορίσω τους ομιλητές για την πρώτη αυτή φάση. Ο Επίτροπος κ. Σαυραμόπουλος θα ξεκινήσει. Ε, θα πρέπει να φύγει στις 9.45 για να παρουσιαστεί στην συνδύση του Κολεγίου των Επιτρόπων. Έχουμε τον προσωπικό ο οποίος εκπροσωπεί την Βουλγαρική Προεδρία, τον Φελίπε ε, Γκονσάλες Μοράλες, ειδικός εισηγητής ε, του ΟΗΕ και κυρία Σαχίν, πρόεδρος ε, του ΚΑΖΙΑΝΤΕΠ, που θα μας παρουσιάσει Πρωτού δώσω το λόγο να αναφερθώ το πώς είναι οργανωμένος ο διάλογος σήμερα Θα δώσουμε ε, το λόγο πρώτα σε δύο μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων και μετά σε ένα μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ώσπου να εξαντληθεί ο κατάλογος των ομιλητών. Μπορεί να φαίνεται περίπλοκο, αλλά θα τα καταφέρουμε. Οι εκπρόσωποι των Εθνικών ε, Κοινοβουλίων που θέλουν να παρέμβουν ε, παρακαλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο και να το παραδώσουν στους κλητήρες. Συμπληρώστε λοιπόν το έντυπο και δώστε το στους κλητήρες. Με βάση αυτά τα έντυπα θα, θα δημιουργηθεί και κατάλογος των μιλητών. Όλοι θα έχουν την ευκαιρία να πάρουν το λόγο. Αυτό με τα οργανωτικά είναι χαρά μου να δώσω το λόγο τώρα στον ε, Επίτροπο, κύριε Βραμμόπουλο, για να ξεκινήσουμε τον πολύ ενδιαφέροντα διάλογο μας. Ευχαριστώ, Κλοντ. Καλημέρα σε όλους. Αγαπητοί συνάδελφοι, υπουργοί, αγαπητή κυρία Δήμαρχε, κύριε Σμετάνοβ, Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να μοιραστώ κάποιε σκέψει σε αυτή την πολύ σημαντική συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Κλοντ, για την πρόσκληση στη σημερινή διακοινοβουλευτική ε, συνεδρίαση για τις νομικές διάβολες και την ένταξη. Ε, εν μέσω μεταναστευτικής και προσφυγικής ε, κρίσης δεν είναι εύκολο να μιλάμε για νόμιμη μετανάστευση και ένταξη. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε την ε, σημασία αυτών των θεμάτων. Μπορεί να μην ε, φαίνονται ως επίγουσες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνουν στο μέλλον. Αν δεν δώσουμε την ε, σωστή προσοχή και αν δεν δράσουμε άμεσα. Η παρουσία όλων σας από όλη την Ευρώπη δεν είναι μόνο επικύρια, αλλά δείχνει ότι Πράγματι έχουμε αυτή τη στιγμή την ευκαιρία την, ε, και την πολιτική στήριξη και την ευθύνη να συζητήσουμε για την νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη. Επενδύοντας την νόμιμη μετανάστευση και στην ένταξη, ε, δεν κάνουμε κάποια φιλανθρωπία, έχει να κάνει με κοινωνική συνοχή, σταθερότητα, έχει σχέση με την οικονομία. Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι και πιο προορατικοί ε, για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να καταρτήσουμε πολιτικές για μετανάστευση στην Ευρώπη. Είναι καιρός να προχωρήσουμε από ε, ένα σύστημα διαχείρισης ε, κρίσης σε μια πιο δομημένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης και να διασφαλίσουμε νομικούς διάβλους να υποστηρίξουμε την ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία. Αυτά όλα αποτελούν τον Ευρωγονέο λίθο για μια τέτοια δομημένη προσέγγιση. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών νόμιμων διόδων γιατί μπορούν άνθρωποι να έρθουν νόμιμοι, νόμιμα στην Ευρώπη για διαφορετικούς ε, λόγους. Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι πώς θα ρυθμίσουμε και θα διχειριστούμε αυτές τις διαφορετικές νομικές προκλήσεις. Η πρόσφατη ε, προσφυγική κρίση μας έδειξε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, να επιτρέπουμε άνθρωποι να ρισκάρουν τις ζωές τους και να ακολουθούν πολύ επικίνδυνες οδούς ε, ο θαλάσσης ή στην ξηρά όταν το μόνο πράγμα που πραγματικά χρειάζεται είναι προστασία. Η επανεγκατάσταση πρέπει, θα πρέπει να είναι προτιμόμενο τρόπος για την ε, παροχή νόμιμων διάβλων. Από το 2015 Θυμόμαστε πώ είχε κατάσταση τότε. Θέλω να σα θυμίσω ότι η Ευρώπη έμεινε έκπληκτη και δεν είχε ιδέα πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση τότε. Το ίδιο ίσχυε φυσικά και για τα κράτη-μέλη. Από τότε λοιπόν Έχουν πραγματοποιηθεί δύο προγράμματα με την κατάσταση και βοήθησαν 26.000 ε, πρόσφυγες να βρουν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα προγράμματα, τα οποία ολοκληρώνονται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε ένα νέο πρόγραμμα ε, το 2017 το Σεπτέμβριο για 50.000 ε, άτομα σε πολύ την κατάσταση ώστε να εισέλθουν μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 40.000 αιτήματα από 19 κράτη-μέλη μέχρι στιγμής. Η Επιτροπή θα παράσχει 500 εκατομμύρια ευρώ ε, μέσα στα επόμενα δύο χρόνια για τη μετεγκατάσταση ε, προσφύγων, 10 ευρώ ε, από τον προϋπολογισμό από κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτείνουμε λοιπόν ένα μόνιμο σχέδιο. Προτείναμε το 2016 τον Ιούλιο ένα μόνιμο σχέδιο για την μετακατάσταση και ορίσαμε μια ενωπημένη ε, διαδικασία και κοινά κριτήρια. Αυτό είναι ένα ε, ουσιαστικό κομμάτι της μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου. Θα δημιουργήσουμε επίσης εναρμονισμένους κανόνες για να διευκολύνουμε, παραδείγματος χάρη, την ε, κοινωνική και οικονομική ένταξη των προσφύγων. Και χωρίς μια συμφωνία και λιγή δεν μπορούμε να έχουμε μια βιώσιμη πολιτική για τη μετανάστευση μακροπρόθεσμα θα εργαστώ ακόμη πιο με τη Βουλγαρική Προεδρία και με τα ε, μέλη του Κοινοβουλίου για να ε, επιτύχουμε μια τέτοια συμφωνία μέχρι τον Ιούνιο και θα ήθελα να συγχαρώ ε, την Βουλγαρική Προεδρία που έχει αναλάβει αυτή τη δέσμευση να επιταχύνει αυτή την διαδικασία. Ταυτόχρονα, και ενώ γνωρίζουμε ότι πάνω από 16 εκατομμύρια άτομα έχουν εκτοπιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο 250 εκατομμύρια βρίσκονται σε κινητικότητα για άλλους λόγους. Ζούμε σε μια εποχή ανθρώπινης κινητικότητας. Έτσι θα μας ε, θα χαρακτηρίσουν αυτή την εποχή ιστορική του μέλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να γίνουμε καλύτεροι στην διαχείριση αυτής της κινητικότητας. Όλοι γνωρίζουμε ότι στο μέλλον η Ευρώπη θα χρειαστεί μετανάστες, γιατί, είναι, γιατί ο πληθυσμός της γυράσκει. Πώς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην υπάρξη εργασιακή δύναμη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί να έλξει ταλέντα από το εξωτερικό για να έχει μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και να ε, ενισχύσει παράλληλα και την ανταγωνιστικότητα. Έχοντας αυτά κατά νου, η Επιτροπή πρότεινε το 2016 την ε, ενίσχυση του προγράμματος ε, της Μπλε Κάρτας. Η έλλειψη δεξιοτήτων και ειδικού εργατικού δυναμικού καταδεικνύει την ανάγκη που, ε, που υπάρχει για να ενισχύσουμε την ε, ελκυστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υψηλά καταρτισμένους ε, εργαζόμενους από το εξωτερικό. Οι μπλε κάρτες και οι εθνικές άδειες για εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ χαμηλότερες από τις άλλες ανταγων... Ε, χώρες ανταγωνιστές όπως, είναι Ευρωπαϊκή... Ε, όπως είναι οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Αυστραλία. Η αναθεώρηση έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις, ε, καθιστώντας το πρόγραμμα πιο ελκυστικό, παράλληλα βελτιώνοντας και ό,τι σχετίζεται με αυτό. Δεν θέλουμε να πούμε στα κράτη-μέλη πόσους ε, ε, ε, εξειδικευμένους εργαζόμενου θα πρέπει να... πώς θα χρειαστούν. Επίσης, δεν θέλω να πούμε στους εργαζόμενους και στις αγορές εργασίας πόσοι ξένοι εργαζόμενοι θα χρειαστούν. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αλλά θέλουμε να κάνουμε το γενικότερο σύστημα πιο ελκυστικό, πιο κινητικό και πιο ευέλικτο. Εκτιμώ ε, ειλικρινά την ε, συνδρομή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του φίλου μου Κλοντ σε αυτό το ε, αντικείμενο. Επίσης, ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια φιλόδοξη, έναν καλό συμβασμό μέχρι τον Ιούνιο και ότι η Βουλγαρική Προεδρία θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε σε αυτό. Η νόμη μετανάστευση δεν έχει όμως να κάνει μόνο με τους υψηλά εξειδικευμένους εργαζόμενους. με ένα ε, έλεγχο καταλληλότητας ε, της ε, νομοθεσίας για την νόμιμη μετανάστευση για το οποίο διαβουλευτήκαμε και με εσά και το οποίο θα ολοκληρωθεί αργότερα αυτό το χρόνο. Είμαι ικανοποιημένο με το ενδιαφέρον που έδειξαν τα ενδιαφερόμενα μέρη. Προς το παρόν αναλύουμε το feedback που έχουμε λάβει η νόμιμη μετανάστευση είναι επίση ένα ε, πολύ σημαντικό συστατικό των ε, σχέσεων μα με τις τρίτες ε, χώρες για την διαχείριση της μετανάστευση. και γι' αυτό τον λόγο συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη για την ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών προγραμμάτων για την μετανάστευση εργασιακού δυναμικού με, συγκεκριμένες, με επιλεγμένες τρίτες χώρες. Τέλος, ένα ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το υποτιμούμε είναι η ένταξη, η κοινωνική και οικονομική ένταξη όλων αυτών που έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον και για τη συνοχή της ε, κοινωνίας μας. Η μεταναστευτική πολιτική και η πολιτική ασύλου μας θα πετύχει μόνο αν η ένταξη των μεταναστών είναι επίσης επιτυχής. Όμως, Χρειαζόμαστε ε, μια νέα προσέγγιση γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο έχουμε εμπλέξει και τον ιδιωτικό τομέα και τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους ε, για να ενισχύσουν και να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους, όπως ε, παραδείγματος χάρη τους εργοδότες, ε, ώστε να δημιουργήσουν εταιρικέ σχέσεις και που θα βοηθήσουν στην ένταξη. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μία ε, ευκαιρία αυτή τη στιγμή. Δεν βρισκόμαστε εκεί που ήμασταν πριν από δύο χρόνια. Η κατάσταση είναι πιο σταθερή και υπό έλεγχο. Πρέπει όμως να είμαστε σε παγρύπνηση. Τώρα πρέπει να δούμε προς το μέλλον και να είμαστε παράλληλα και φιλόδοξοι και έξυπνοι, σχεδιάζοντας μια μεταναστευτική πολιτική ε, που θα εντέξει στο μέλλον να ενισχύσουμε την νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη ε, γιατί αυτά τα δύο είναι, τα, ε, είναι βασικά κομμάτια ενό ε, μεγαλύτερου πάζλου. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μοιραστώ τη σκέψη μου μαζί σα και σας εύχομαι μια επικοδομητική συζήτηση σήμερα και βασίζομαι επίση στην υποστήριξή σας για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Commissioner. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ξέρω ότι θα αποχωρήσετε για να μεταβείτε στην συνεδρίαση της Επιτροπής, των Επιτρόπων συγκεκριμένα. Όμως είμαστε πάντα σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα τα όσα ακούσαμε από εσά. Και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Μπέρνερ. Αναπληρωτή Υπουργό Ιστορικών που εκπροσωπεί τη Βουλγαρική Προεδρία. Οι προσεχείς μήνες ξέρουμε ότι θα είναι, θα είναι γεμάτοι προκλήσεις από τα πιο ε, πλήρη πακέτα δουλειάς ε, από το μεγαλύτερο κομμάτι της ε, δουλειάς και βέβαια με τομείς πολύ ευαίσθητους θα πρέπει εσείς να ολοκληρώσετε και να φέρετε εις πέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ και εσάς για την παρουσία σας και σας δίνουμε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Σβετάνο. Αξιότιμη κύριε Επίτροπε, κύριε Αβραμόπουλε, Αξιότιμη κυρίες και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκληση αυτή, για συμμετοχή στην ε, διακοινοβουλευτική συνεδρίαση της Επιτροπής σας. Είναι τιμή για μένα το ότι μπορώ να εκπροσωπήσω την Προεδρία την Βουλγαρική Προεδρία. Βεβαίως ε, το θέμα της ε, μετανάστευσης και οι διαδικασίες ε, μακροπρόθεσμα έχουν ε, προσελκύσει το ενδιαφέρον και την επικαιρότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι μια ολιστική διαχείριση της μετανάστευσης θα απαιτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποφασιστική δράση και για την αντιμετώπιση της παράνομης, της παράτοπης, της λαθρέας διακίνησης, τη συνεργασία με τρίτες χώρες, με διεθνείς οργανισμούς. Είναι ένα πολύ σχεδέ ζήτημα δηλαδή και η Βουλγαρική Προεδρία είναι διατεθειμένη να συνεχίσει και να ε, παγιώσει, να τις προσπάθειες για τη βελτίωση της αντιμετώπισης των προβλημάτων των σχετικών με τη μετανάστευση και για την εξασφάλιση μιας ολιστικής διαχείρισης με την εσωτερική αλλά και εξωτερική διάσταση μιας ε, πολιτικής δηλαδή καλά ισορροπημένη σε σχέση με το μεταναστευτικό φαινόμενο. Θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας και σταδιακά θα ε, μετατοπιστεί πιστεύουμε το ενδιαφέρον από την ανάγκη για διαχείριση μιας κρίσης μεταναστευτικής σε μια διαχείριση μακροπρόθεσμη, σε μια προσέγγιση μακροπρόθεσμη στην μεταλλαγή των έκτακτων και παράτυπων μεταναστευτικών ροών σε σχεδιασμένες και νόμιμες ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξουμε ότι δεν είναι δυνατόν να διαμένουν παράνομα στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, άνθρωποι που έχουν μπει χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις, ενώ ταυτόχρονα δεν υπάρχει η δυνατότητα για ε, οργανωμένες και νόμες μεταναστευτικές πολιτικές. Αυτό πρέπει να το δείξουμε σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε ως Βουλγαρική Προεδρία όλες τις προσπάθειες για μόνιμες και αποτελεσματικές ε, λύσεις συνεργασίας με όλους τους εμπλεκομένους. Βεβαίως ε, είμαστε εν γνώση των φαινομένων των δημογραφικών που αφορούν τα κράτη-μέλη και που μας οδηγούν όπως οι δημογραφικές αλλαγές, όπως η γύρανση του πληθυσμού ε, και τα προβλήματα που αυτά συνεπάγονται και που μπορούμε πιστεύουμε να λύσουμε χάρη σε μια καλή μεταναστευτική πολιτική, προσέλκυση ανθρώπων με υψηλές δεξιότητες ε, και οργάνωση μιας καλής αγοράς εργασίας στα κράτη-μέλη. Μπορούμε λοιπόν σε συνεργασία οι συνομοθέτες σε σχέση με ορισμένα διφλονικούμενα ζητήματα, με κάποια ακόμη επίμαχα σου ζητήματα όπως είναι η μπλε κάρτα, να βρούμε λύσεις, να βρούμε κοινά οράματα για την οργάνωση για τη βελτίωση της ελκυστικότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης για ε, υπηκόους τρίτων κρατών με υψηλά προσόντα και δεξιότητες, για βελτίωση των συνθήκων στην αγορά εργασίας και βεβαίως για εξασφάλιση συνθήκων τέτοιων για τους υπηκόους των τρίτων χωρών, ώστε και ευχερέστερα να εξασφαλίζεται η κινητικότητά τους, αλλά και να ε, είναι πιο ευχερής για αυτούς η απόφαση να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέσα λοιπόν για την μετανάστευση, η θεώρηση διαβατηρίων για τους φοιτητές παραδείγματι, η περιστασιακή, η εποχιακή εργασία ε, μπορεί να προσελκύσει ε, μπορούν να προσελκύσουν ανθρώπους ικανούς με προσόντα σε θέσεις εργασίας που έχουν υψηλές απαιτήσει και αυτό μπορεί να συμβάλλει και στην ε, οργάνωση της μεταναστευτικής πολιτικής γενικότερα χάρη σε ένα σχέδιο μετεγκατάστασης ε, το οποίο θα λειτουργεί ικανοποιητικά και για αυτούς που χρειάζονται προστασία σε όρους διασφάλισης των δικαιωμάτων βέβαια και της αξιοπρέπειάς τους. Χρειάζεται ένα νόμιμο πλαίσιο όμως. Και αυτό πρέπει να προαχθεί σε όρους ανθρωπιστικούς, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι όροι υποδοχής εκείνων που έχουν ανάγκη προστασίας σε όρους εθελοντικούς για τα κράτη-μέλη μέσα από προγράμματα μετεγκατάστασης εθνικά με ταυτόχρονη διασφάλιση και της ασφάλειας για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς όμως να επιτρέπεται καμία κατάχρηση δικαιωμάτων χωρίς να παραβιάζονται οι εγγύησεις των δικαιωμάτων που ε, προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επανεξετάσουμε τι μέτρα προβλέφθηκαν από το 2007 μέχρι τώρα για την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης της μετανάστευσης και να τα καθοδηγήσουμε προς συγκεκριμένα και καλύτερα αποτελέσματα, μηχανισμούς θεώρησης διαβατηρίων, παραδείγματι, και άλλους μηχανισμούς που μπορούν να οδηγήσουν σε μία προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από θεώρηση, υποχρέωση θεώρηση διαβατηρίων σε περίπτωση όπου είναι οι συνθήκες ασφάλειας ή οι μεταναστευτικές συνθήκες ε, πιεστικές ή έκτακτες ή απειλητικές για ένα κράτος. Ε, συστήματα λοιπόν που θα πρέπει να εξετάσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες πάντα σε αναζήτηση της λεπτής ισορροπίας μεταξύ της διευκόλυνσης βεβαίως των ε, ε ταξιδίων ε, και ενός συστήματος θεώρησης διαβατηρίων αλλά και ταυτόχρονα της προστασίας των κρατών μας. Εξετάζουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να προχωρήσουμε προς μια μεγαλύτερη εναρμόνιση της πολιτικής για τη θεώρηση των διαβατηρίων. Είμαστε διατεθειμένοι να αρχίσουμε την ε, επεξεργασία των τροπολογιών για τον κώδικα για την θεώρηση διαβατηρίων και το σύστημα ρύθμισης των θεωρήσεων και ε, μπορούμε χάρη σε αυτά πιστεύουμε να ενισχύσουμε τη διαχείριση και τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως Προεδρία εμείς θα ασχοληθούμε με την ουσία των ε, ροών ε, και της πολιτικής για τη μετανάστευση στο σύνολο των προτάσεων, το πακέτο δηλαδή για τη μετανάστευση με την ε, βούληση να ενισχύσουμε την ε, ρύθμιση της μετανάστευσης των μεταναστευτικών ροών σε συνεργασία ασφαλώς με τις χώρες προελεύσεως, με δυνατότητες για ε, επανένταξη στην αγορά εργασίας όσων επαναπατρίζονται, σε συνεργασία τους από τις χώρες προελεύσεως και με τις χώρες διελεύσεως και πρέπει ιδιαίτερα να στραφούμε στην αντιμετώπιση των αιτίων της μετανάστευσης. Αυτό θα το εξασφαλίσουμε με, την, ε, με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη για το 2020. Η συνεργασία θα είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ολιστικής προσέγγισης για τη μετανάστευση. Πιστεύουμε σε μια στενή συνεργασία, σε ανοιχτό και ρεαλιστικό πραγματιστικό διάλογο με τις χώρες προελεύσεως και διελεύσεως. Ε, με το πρόγραμμα δράσεως για τη Βαλέτα έχουμε σημαντικά εργαλεία, όπως και με το πρόγραμμα εταιρική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με συγκεκριμένα προγράμματα συνεργασίας με τρίτες χώρες, που μπορούν να αναπτυχθούν για να φέρουν πλήρη αποτελέσματα. Πιστεύουμε στη συνεργασία στο πλαίσιο εταιρικών σχέσεων με υποστήριξη και βελτίωση των δυνατοτήτων μας για καλύτερη διαχείριση της μετανάστευσης ε, και μια προσέγγιση που θα πρέπει να αποβεί εποφελής για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των περιφερειών, ιδιαίτερα εκείνων που πλήττονται περισσότερο από την φτώχεια, πρέπει να αντιμετωπιστεί στο, με τον τρόπο αυτό η ρίζα του κακού, η, τα αίτια δηλαδή της μετανάστευσης και πρέπει να στραφούμε και προς τις χώρες, ε, τις τρίτες χώρες που είναι έτοιμες να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους δίνουμε χείρα εφόσον είναι διατεθειμένες να βελτιώσουν τις δυνατότητες τους για ε, επανυποδοχή των παρατύπων μεταναστών και την επανένταξή τους. Πρέπει να έχουμε μια στρατηγική προσέγγιση ε, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουμε την αιτία της στρατηγικής, των στρατηγικών μεταναστευτικών ρόλων, της στρατηγικής εκδοχής του φαινομένου. Επίσης πρέπει να έχουμε συστήματα διευκόλυνσης της θεώρησης για να διευκολύνεται η νόμιμη μετανάστευση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα συμβάλλει στην βελτίωση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες στον τομέα της νόμιμης πρόσβασης. Θα βελτιώσει την αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μειώσει τις ε, παράτυπες ροές. Η Βουλγαρική Προεδρία είναι διατεθειμένη να συμβάλλει στο μέτρο των δυναμεών της ε, στην ε, ενίσχυση των νόμιμων ροών που θα πρέπει να αποτελέσουν μια πραγματική εναλλακτική σε σχέση με την παράνομη διέλευση των συνόρων. Και έτσι θα καμφθούν όλα τα φαινόμενα και κυρίως ε, οι μεγάλη κίνδυνοι και οι προκλήσεις που σημαίνει η παρανομετανάστευση. μετανάστευση. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε με τους ε, συντέρους μας στις άλλες χώρες να κάμψουμε ε, εισάγοντας νόμιμες οδούς τις δυσμενείς συνέπειες αυτής της του των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Θερμό καλωσόρισμα. δεν λειτουργεί το μικρόφωνο του κύριου Μοράλες. Σας ευχαριστώ. Ε, τον περασμένο Αύγουστο ανέλαβα τα καθήκοντά μου και κατά τη θητεία μου θα προσπαθήσω να ενισχύσω τα δικαι... την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ε, μεταναστών ε, που συνήθως είναι ευάλωτοι και αφανείς. Ε, δεν πρέπει να θεωρούμε τη μετανάστευση πρόβλημα, ούτε και τους μετανάστες πρόβλημα. Διαφορετικά βέβαια είναι τα προβλήματα που μπορούν να ανακύψουν εξαιτία ακατάλληλων πολιτικών και πρακτικών των κρατών μελών. Το διακύβευμα εδώ είναι πώς τα κράτη αντιμετωπίζουν τη μετανάστευση. Ε, μετανάστευση υπήρχε ανέκαθεν και θα υπάρχει πάντα. Ε, είναι ε, χαρακτηριστικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς να αναζητεί καλύτερες ευκαιρίες ε, για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Και πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις των μεταναστών για το πότε, γιατί, πού και με ποιο τρόπο θα μεταναστεύσουν. Και βασικοί παράγοντε που του εξωθούν στη μετανάστευση είναι η φτώχεια, η βία, η διάκριση, η κακή διακυβέρνηση. Ενώ οι ε, βασικοί παράγοντε που του έλκουν προ μια χώρα είναι επίσημε ή μη αναγνωρισμένε εργασιακέ ανάγκε και επανένωση οικογενειακή. Ε, Κυρίω πηγαίνουν οι μετανάστε εκεί που υπάρχουν δουλειέ, που μπορούν να ενταχθούν κοινωνικά και να δημιουργήσουν ένα μέλλον για τα παιδιά του. Και μάλιστα η δημόσια συζήτηση μερικές φορές παρά είναι ρηχή και καθιστά από διαπομπέους τράγους τους ε, μετανάστες. Ε, κατηγορώντας ότι τους κλέβουν τους δουλειά. Η δημόσια συζήτηση μερικές φορές παρά είναι ρηχή και καθιστά από διαπομπέους τράγους τους ε, μετανάστες. κατηγορώντα ότι του κλέβουν τους δουλειά. Κυρίως δουλειά στην Ήπεθρο, στη Γεωργία, στι οικοδομέ φιλοξενία, εξόριξη, αλληλεία και πολλές φορές είναι θύματα ταχύ πόδι του σε άλλη χώρα μπαίνουν στον κίνδυνο να παίξουν τη ζωή του κορώνα γράμματα για να το πετύχουν. Και μάλιστα μερικέ φορέ κάνουν τι βρώμικε δουλειέ, τι πιο επικίνδυνε και τι δύσκολε τη οικονομία των ε, χωρών του Παγκόσμιου Βορρά. Μάλιστα, οι δημογραφικέ αλλαγέ και η γύρωση του πληθυσμού θα πρέπει να οδηγήσει σε νέου τρόπου αντίληψη τη μετανάστευση. Και όλοι οι μετανάστε αξίζουν ε, προσιτές, ε, ε, νόμιμες, ασφαλείς και προσβάσιμες διόδους για να μεταναστεύσουν και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίες. Οι κατασταλτικές πολιτικές και έλλειψη απαντήσεων για, τους, για τα αίτητρο διακίνησης. Γιατί τα κράτη-μέλη δεν αντιμετωπίζουν τα αίτια ε, της μετανάστευση και η λεγόμενη μεταναστευτική κρίση είναι κυρίω κρίση πολιτικής βούληση και η δημιουργία περιορισμών των μεταναστευτικών κινήσεων είναι τμήμα του προβλήματο και όχι μέρος της λύσης. Πολιτικές αποτροπής όπως ιστότους ε, της οικογενειακής επανένωσης απλώς ε, επιτείνουν τα δεινά και το, το τραύμα, το ψυχολογικό που υφίστανται οι μετανάστες και υποσκάπτουν την ένταξή τους. Και ο προκατοχός μου και εγώ έχουμε επισημάνει επανειλημμένως ε, τις ανησυχίες μας για την ε, δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας και τη συμφωνία με την ε, Λιβύη, γιατί ίσως έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραβιάζει τι διεθνεί και των σύνορων, προκειμένου να μείνουν, παραμείνουν όσο πιο μακριά γίνεται από τα εξωτερικά σύνορα οι μετανάστες και οι οδύνες τους, η ταλαιπωρία τους και τα δεινά τους και με πιο νόμιμους, ε, προσιτούς ε, και ασφαλείς ε, διάβλους θα εξασφαλίσουμε καλύτερη θέση των μεταναστών προκειμένου να... η μετανάστευση στηρίζει την ανάπτυξη και την ευημερία και έχει γενικό θετικό αντίκτυπο στη δημιουργία θέσεων απασχόληση και σε επενδύσει. Οι μετανάστε συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη όπου και ποιε που ευνοούν την ε, πολυμορφία και την ένταξη των ε, μεταναστών περιορίζοντας ε, λαϊκιστικές δοντών τους. Θα πρέπει να υιοθετήσουμε πολιτικές που δεν θα ευκολύνουν τη μετακίνηση και θα δίνουν στους, στα κράτη, στα κράτη τη, το εργατική επανένωση άδεια εργασίας ή βίζα εργασίας διαμένοντος θεώρηση σύνταξης ή φοιτητική θεώρηση με όλους τους απαραίτητους Γιατί ε, οι μετανάστες δεν θέλουν να παραμείνουν χωρίς χαρτιά, να χρησιμοποιήσουν λαθροδιακινητές. Είναι λύση απελπισίας και θα προτιμούσαν κάλλιστα να πληρώσουν ε, ένα λογικό τέλος σε έναν ε, υπεύθυνο θεωρήσεων παρά να υποφέρουν τον εκβιασμό των λαθροδιακινητών και θα προσαρμοστούν στις απαιτήσει των κρατών για να έχουν πρόσβαση στην νόμιμη κινητικότητα και προτιμούν να ε, ενταχθούν σε ένα σύστημα με κανονικά ταξιδιωτικά έξοδα από την υποστούν την ταλαιπωρία ενό αβέβαιου ταξιδιού. Και μάλιστα θα προτιμούσαν μια επίσημη αγορά εργασία Και ε, σίγουρα ο καλύτερος ε, στόχος της διαχείρισης της κινητικότητας είναι η προσφορά νόμιμων διάβλων. Έτσι θα περιορίσουμε την λαθραγορά της λαθροδιακίνησης και Ίσως θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι τα προέλευσης, ενώ ε, υπάρχουν αντίστοιχες προ... ευκαιρίες στις χώρες υποδοχής. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις ε, ανάγκες και των αγορών εργασίας και να δώσουμε ε, λύσεις στους μετανάστες και να μην τους αφήσουμε θύματα αδίστακτων λαθροδιακινητών και σπυρών. Φυσικά θα περιορίσει την ισχύ των λαθροδιακινητών και η δυνατότητα πρόσβαση στην επίσημη αγορά εργασία θα δημιουργήσει ευκαιρίε και για του εργαζόμενου και για του εργοδότε. Η κατάργηση των προσωρινών προγραμμάτων απασχόληση ε, μεταναστών βάσει χορηγίε και οι ανοιχτέ ε, ε, θεωρήσει εργασία, θεωρήσεων ανθρωπιστικών και άλλων ευκαιριών, τα κράτη-μέλη θα μπορέσουν να αναπτύξουν κατάλληλου μηχανισμού για την επανεγκατάσταση των προσφύγων. Θέλουμε τέτοια καλή διαχείριση των προγραμμάτων και τέτοιου είδου προγράμματα με ανθρωπιστικέ θεωρήσει θα δημιουργήσουν ευκαιρίε για ένα μακροπρόθεσμο αξιόπιστο πρόγραμμα ώστε ένα μεγάλο αριθμό των προσφύγων να επιδιώξει την επανεγκατάσταση αντί να ε, ξοδεύει ε, υπέρογκα ποσά και να παίζει τη ζωή του κοροναγράμματα στα χέρια των λαθροδιακίνητων. Και αυτό θα μειώσει και την αγορά για τους λαθροδιακίνητες και το κόστος ε, της διαδικασίας της αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα. Όπως είπα, οι λαθραγορές εργασίας είναι μαγνήτης ε, για την παράτυπη μετανάστευση και είναι ο βασικός κανόνας ε, και παράγων ε, προσέλκυσης των μεταναστών και έναυσμα των, της λαθραγοράς εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να μειώσουμε αυτές τις λαθραγορές ή μη θα έχουμε αρνητικές συνέπειες σε πολλούς τομείς. Για παράδειγμα, στις οικοδομές, στη γεωργία, στη φιλοξενία, ε, τη φροντίδα, τις εξορίξεις, ε, με τη συγκατάθεση μερικές φορές των καταναλωτών, την αδιαφορία των πολιτικών και την έλλειψη ε, προσφυγών των μεταναστών φοβούμενων την, ε, την κράτηση, την κράτηση, τη σύλληψη, ε, δυστυχώς συνεχίζονται τι πρακτικές. Θα πρέπει να αποφύγουμε επίση στρέβλωση της αγοράς εργασίας ε, με κατάλληλου ε, μηχανισμού εργασιακή επιθεώρησης με στόχο τους εκμεταλλευτές εργοδότε, προκειμένου να ενισχύσουμε τα δικαιώματα των μεταναστών. Κάποιε προορατικέ διαδικασίε νομιμοποίηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμε και να βοηθούν του εργαζόμενους μετανάστες να ενταχθούν κοινωνικά με κατάλληλο νομικό καθεστώς για να καταπολεμήσουμε την εκμετάλλευση και να προασπίσουμε τα δικαιώματά τους που είναι δικαιώματα και των υπόλοιπων εργαζομένων. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ πολύ. Πρωτού προχωρήσω στον τελευταίο μιλητή. Έχω να κάνω μια συνήθιτη ανακοίνωση. Κάποιος έχει αφήσει ένα δαχτυλίδι πολύτιμο στο αν ανοίξει κάποιον από εσά. Ε, να μας το πείτε στο τέλος της συνεδρίασης και θα σας επιστραφεί. Ε, δεν αστιεύομαι, όντως. Θα το επιστρέψουμε διακριτικά. Δεν θα σχολιάσω άλλο. Σουρεαλιστική ανακοίνωση. Αγαπητοί συνάδελφοι, αν γνωρίζω ότι κάποιοι από εσά έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία σε θέματα ένταξης στα κρατημέλη και στις περιφέρειες. Η επόμενη μας ομιλήτρια θα μιλήσει για αυτό το θέμα ακριβώ, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία. Είναι η Δήμαρχος Φάτμα Σαχίν και θα ήθελα να, να πω σε αυτούς που δεν έχουν πάει στην Καζάντιεπ στην Τουρκία ότι είναι μια επαρχία η οποία το 2016 προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης για τον τρόπο που υποδέχτηκε τους ε, Σύριους πρόσφυγε σε μικρό χρονικό διάστημα, σε σύντομο χρονικό διάστημα δέχτηκε 50.000 ε, πρόσφυγες έχει βοηθήσει στην κατάσταση διπλασίου αριθμού ε, ατόμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε σίγουρα η κυρία Σαχίν ξέρει πώς μπο, ε, μπορεί να έχει βοηθήσει στην κατάσταση διπλασίου αριθμού ε, ατόμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία δύο χρόνια. Οπότε σίγουρα η κυρία Σαχίν ξέρει πώς μπο, ε, μπορεί να μας βοηθήσει με την εμπειρία της. Της δίνω λοιπόν το λόγο για να μας μιλήσει για την εμπειρία αυτή. Κυρία Σαχίν. Sayın Başkan, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, όπως είπε και ο κύριο Πρόεδρος σήμερα, συζητούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα και θέλω να σας παρουσιάσω ένα πολύ σημαντικό και αναγνωρισμένο ανά τον κόσμο μοντέλο υποδοχής όπως αυτό του ΑΝΤΕΠ, του Γκαζιαντέπ. Ήθελα λοιπόν να σας, δω πώς, να σας πω πώς ε, υποδεχθήκαμε, πώς αντιμετωπίσαμε το φαινόμενο της μετανάστευσης στο Γκαζιάντσεπ. Να σας παρουσιάσω όμως πρώτα την ε, πόλη. Είναι στον ε, κατάλογο της UNESCO για τις πόλεις με αρχαίους πολιτισμούς στα προστατευμένα δηλαδή, στις πόλεις που τίθενται υπό την προστασία της UNESCO. Αυτή είναι η πόλη της οποίας είμαι δήμαρχος, στον Καζιάντεπ. Από το 2010 και μετά ε, που αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα ε, μας απασχόλησε το πώς μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα προβλήματα και ξέρετε ότι εμείς και η τουρκική κυβέρνηση με πρώτο γνώμονα και μέλημα την ανθρωπιά την ανθρώπινη προσέγγιση και την ενσυναίσθηση προς τον συνάνθρωπο κάναμε προσπάθειες για να δώσουμε απάντηση στα προβλήματα. Όπως είπε και ο κύριος ε, Πρόεδρος νωρίτερα, ήταν πολύ μεγάλο το βάρος ε, των μεταναστευτικών ροών που αντιμετώπισε η Τουρκία και περιοχή μας, ειδικότερα πολύ μεγαλύτερο από ότι οπουδήποτε αλλού, οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου. Βέβαια, το σηκώσαμε το βάρος και θέλω να σας εξηγήσω πώς τα καταφέραμε. Το μεγαλύτερο μάλιστα βάρος μεταναστευτικών όρων ε, το έχει σηκώσει η δική μου υπόλοιπη περιοχή μας. Με την συμφωνία που συνήφθη με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίστηκε βεβαίως ότι είναι τεράστια η πίεση και ότι πρέπει να μειωθούν οι αριθμοί. Και αυτό πρέπει να σας το εξηγήσω γιατί έγιναν αυτές, γιατί δόθηκαν αυτές οι λύσεις. Ε, πρέπει να σας εξηγήσω πόσο αφόρητα ήταν η πίεση ε, και ότι αυτό ήταν ο καταγγελότερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τι έκανε λοιπόν το Αντέπ, το Γκαζί Αντέπ. Ξέρετε ότι εγώ ήμουν πριν πρόεδρο, ε, υπουργός ε, οικογένειας και βέβαια από ε, τα καθήκοντά μου αυτά ήδη είχα βρεθεί αντιμέτωπη με τα θέματα της ε, μετανάστευσης. Είχα ασχοληθεί με τη μέσο και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση και το σχεδιασμό. Κύριο μέλημά μας λοιπόν και καταλάβαμε ότι αυτό είναι και η λύση ήταν η από κοινού διαχείριση, η από κοινού αντιμετώπιση. Φερρυπίν, μπορεί εμείς στην ε, ε, περιοχή μας να χρειάστηκε να ανοίξουμε σχολεία γιατί είχαμε παιδιά ορφανά από πατέρα και μητέρα που είχαν φτάσει στην περιοχή μας, στην πόλη μας, στον Καζιαντέπ και δεν είχαν σχολείο να πάνε και θα πέφτανε στα χέρια μιας τρομοκρατικής οργάνωσης ή του Ισλαμικού κράτους ή του ΠΚΚ. Και έτσι έπρεπε να μεριμνήσουμε για σχολεία. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε εδώ και 7 χρόνια ως ε, ε, μητροπολιτική ζώνη του Γκαζιαντέπ. Ανοίξαμε μάλιστα και ένα κέντρο ε, το οποίο για να το ανοίξουμε κάναμε την έρευνα. Τι χρειάζεται, τι χρειάζεται μια κοινωνία ή μια κοινωνική ομάδα για να μπορέσει να ενταχθεί στην κοινωνία υποδοχής. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια πιο αρμονική συμβίωση. Κάναμε λοιπόν την έρευνα πρώτα για να ανοίξουμε το κέντρο αυτό που εξυπηρετεί τις κοινωνικές πολιτικές. Με μια σειρά από μαθήματα που προσφέρουμε σε γυναίκες, πρόσφυγες, σε παιδιά, για να αποτρέψουμε την γετοποίηση. Γετοποίηση η οποία οπωσδήποτε έχει σαν επόμενο βήμα την ε, ρίζοσπαστικοποίηση. Αυτός ήταν ε, ο γνώμονας με τον οποίο προχωρήσαμε. Προσφέραμε μαθήματα γλώσσας, προσφέραμε μαθήματα ε, επαγγελματικής κατάρτισης και πάνω απ' όλα θελήσαμε να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανθρωπιά, την δυνατότητα να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Και βεβαίως Πρώτος στόχος μας ήταν να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά, γιατί έχουμε αυτήν την θεμελιώδη ε, φιλοσοφική προσέγγιση που άλλωστε είναι κοινή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γυναίκα, το παιδί πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη φροντίδα και περιποίηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε με την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουμε σε ταχύτερη ε, εξασφάλιση των αναγκών ε, και της υποστήριξης που χρειάζεται, μέχρι και παιδικούς σταθμούς, σε παραδείγμα την μπορέσαμε να ανοίξουμε και διατηρούμε. Το Gaziantep, ε, για να σας δώσω μια εικόνα σε αδρές γραμμές, υποδέχτηκε μέσα στην τελευταία επταετία πληθυσμό μεταναστών και προσφύγων ισοδύναμο με αυτό, τον Βρυξελ, το, με το, με αυτό του 50% του πληθυσμού των Βρυξελών. Καταλαβαίνετε τι σήμαινε αυτό και σε όρους ε, παρεχόμενης στέγης και λοιπόν υποδομών. 17.000 μόνο είναι τα παιδιά τα οποία είναι ε, ανήλικα και υποδεχόμαστε κάτω από 18 ετών δηλαδή με σχολεία τα οποία έχουμε προσφέρει εμείς, τα οποία έχουμε οργανώσει ε, κατά τρόπον ώστε το 67% τουλάχιστον των παιδιών ε, μπόρεσαν να ε, μπουν στο σχολείο μέσα στην πρώτη τετραετία από την, άφηξη, από την εκκίνηση του φαινομένου αυτού. Πρέπει να σας πω ότι τα ποσοστά τα οποία έχουμε επιτύχει, τα ποσοστά προσφοράς παιδείας και εκπαίδευση στα παιδιά αυτά είναι ισοδύναμα με αυτά που θα είχαν, αν όχι καλύτερα, με αυτά που θα είχαν στην στην πατρίδα. Αν είχαν μείνει στη Συρία δηλαδή, θα είχαν τα ίδια ποσοστά ε, ε παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο. Το ίδιο σε σχέση και με την εργασία και απασχόληση. Έχουμε ξεκινήσει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την εξασφάλιση θέσεως εργασίας χωρίς ποσοστώσεις, χωρίς αποκλεισμούς στους υποψηφίους εργαζομένους. Και έτσι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό ε, πρόγραμμα. Έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο πρόγραμμα επίσης με ε, κανάλια αρδευτικά, 120 χιλιόμετρα συνολικά, ε, το οποίο εξασφαλίζει την ίδρευση, την άρδευση και γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι μιλούμε για ένα συνολικό μοντέλο του Γκαζιάντεπ. Είδατε πόσο πυλισχυδές είναι αυτό. Ουσιαστικά χρειάστηκε να χτίσουμε μια καινούργια πόλη. Γιατί, Γιατί έφτανε πολύ ε, υψηλά το ενίκιο στα υφιστάμενα, στην υφιστάμενη στέγη, καθώς υπάρχει και ε, παρουσία στρατιωτική στην περιοχή και άρα ε, αυτό ούτως ή άλλως ε, πίεζε προς τα πάνω τα ενίκια. Χρειάστηκε λοιπόν να φτιάξουμε καινούρια στέγη, να χτίσουμε καινούριες κατοικίες. Εμείς, για να σας εξηγήσω την προσέγγιση μας, την μετανάστευση την είδαμε σαν ένα αποτέλεσμα, όχι σαν ένα αίτιο. Ότι δηλαδή, εάν υπάρχουν αυτές και αυτές οι συνθήκες, τότε υπάρχει πίεση μεταναστευτική. για οποιονδήποτε μπορεί να διαμαρτύρεται για τη μετανάστευση, θα συνιστούσα να κοιτάξει ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους κάποιος άνθρωπος αφήνει το σπίτι του και μεταναστεύει. Κοιτάξτε τη Μέση Ανατολή όχι ως μια πηγή πετρελαϊκών πόρων, όχι ως ένα διάβλο των μεγάλων αγωγών του πετρελαίου. Κοιτάξτε την σαν μια πηγή ε, ανθρώπων ε, με δυνατότητες που έχουν ανάγκη από ενσωμάτωση στις κοινωνίες, που μπορούν να αποτελέσουν το για όλες τις κοινωνίες, όπως αποδείχθηκε και για τον Καζίαν Τεπ. Η συζήτηση ε, που κάνουμε σήμερα ε, είναι πολύ σημαντική και γιατί μας επιτρέπει να ε, μιλήσουμε για τον Gaziantep, για τα προγράμματα, τα εθελοντικά που αναπτύχθηκαν, αλλά ταυτόχρονα τονίσουμε και το γεγονός ότι η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτική σημασία για μας γιατί εξασφαλίζει μια σταθερότητα στις ροές Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούστηκε νωρίτερα ότι πρέπει να ε, δοθούν δυνατότητες για νόμισμη μετανάστευση. Πρέπει η μετανάστευση όμως να δώσει δυνατότητες όχι μόνο σε αυτόν που είναι εποφελής ή χρήσιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δώσει δυνατότητες και, στον, ε, και στο παιδί, το ορφανό, τον ηλικιωμένο, τον άρρωστο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί ανθρωπιά από τον κόσμο. Αυτή είναι η δική μου η έκκληση ε, η δική μου έκκληση, σας μιλώ ως γυναίκα, σας μιλώ ως άνθρωπος, να ανοίξουμε τις αγκαλιές μας, να δείξουμε μια πιο ανθρώπινη, ε, ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει την αγκαλιά της και να υποδεχθεί περισσότερους ανθρώπους. Αυτά ήθελα να σας πω για το μοντέλο του Γκαζιαντέπ, να μοιραστώ μαζί σας και κυρίω να μιλήσω για την ανθρωπιά, για το δίκαιο του ορφανού, για το δίκαιο της γυναίκας, για το δίκαιο του ηλικιωμένου. Και ελπίζω, ελπίζω και πιστεύω ότι πρέπει να αναλυφθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε κάθε περιοχή του κόσμου. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε κυρία Δήμαρχε Σαχίν. Σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσετε την εμπειρία αυτή. Κυρία Σαχίν. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κυρίες και κύριοι, όπως είπε και ο Πρόεδρος σήμερα, συζητούμε ένα πολύ σημαντικό θέμα και θέλω να σας παρουσιάσω ένα πολύ σημαντικό και αναγνωρισμένο ανά τον κόσμο μοντέλο υποδοχής όπως αυτό του ΑΝΤΕΠ, του Γκαζιαντέπ. Θέλω λοιπόν να σας, δω πώς, να σας πω πώς ε, υποδεχθήκαμε, πώς αντιμετωπίσαμε το φαινόμενο της μετανάστευσης στο Γκαζιαντέπ. Να σας παρουσιάσω όμως πρώτα την ε, πόλη είναι στον κατάλογο της UNESCO ε, για τις πόλεις με αρχαίους πολιτισμούς, στα προστατευμένα δηλαδή, στις πόλεις που τίθενται υπό την προστασία της UNESCO. Αυτή είναι η πόλη της οποίας είμαι δήμαρχος, στον Καζιάντεπ. Από το 2010 και μετά ε, που αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε τα φαινόμενα ε, μας απασχόλησε το πώς μπορούμε να δώσουμε απάντηση στα προβλήματα και ξέρετε ότι εμείς και η τουρκική κυβέρνηση με πρώτο γνώμονα και μέλημα την ανθρωπιά την ανθρώπινη προσέγγιση και την ενσυναίσθηση προς τον συνάνθρωπο κάναμε προσπάθειες για να δώσουμε απάντηση στα προβλήματα. Όπως είπε και ο κύριος ε, Πρόεδρος νωρίτερα, ήταν πολύ μεγάλο το βάρος ε, των μεταναστευτικών ροών που αντιμετώπισε η Τουρκία και η περιοχή μας, ειδικότερα πολύ μεγαλύτερο από ότι οπουδήποτε αλλού, οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου. Βέβαια, το σηκώσαμε το βάρος και θέλω να σας εξηγήσω πώς τα καταφέραμε. Το μεγαλύτερο μάλιστα βάρος μεταναστευτικών όρων ε, το έχει σηκώσει η δική μου η περιοχή μας. Με την συμφωνία που συνήφθη με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίστηκε βεβαίως ότι είναι τεράστια η πίεση και ότι πρέπει να μειωθούν οι αριθμοί και αυτό πρέπει να σας το εξηγήσω γιατί έγιναν αυτές, γιατί δόθηκαν αυτές οι λύσεις. Ε, πρέπει να σας εξηγήσω πόσο αφόρητα ήταν η πίεση ε, και ότι αυτό ήταν ο καταλληλότερος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Τι έκανε λοιπόν το ΑΝΤΕΠ, το Γκαζί ΑΝΤΕΠ. Ξέρετε ότι εγώ ήμουν πριν πρόεδρο, ε, υπουργός ε, οικογένειας και βέβαια από ε, τα καθήκοντά μου αυτά ήδη είχα βρεθεί αντιμέτωπη με τα θέματα της ε, μετανάστευσης. Είχα ασχοληθεί με τη μέσο και προθεσμή αντιμετώπιση και το σχεδιασμό. Κύριο μέλημά μας λοιπόν και καταλάβαμε ότι αυτό είναι και η λύση ήταν η από κοινού διαχείριση, η από κοινού αντιμετώπιση. Φερρυπίν, μπορεί εμείς στην ε, ε, περιοχή μας να χρειάστηκε να ανοίξουμε σχολεία γιατί είχαμε παιδιά ορφανά από πατέρα και μητέρα που είχαν φτάσει στην περιοχή μας, στην πόλη μας, στον Καζιαντέπ και δεν είχαν σχολείο να πάνε και θα πέφτανε στα χέρια μιας τρομοκρατικής οργάνωσης ή του Ισλαμικού κράτους ή του ΠΚΚ. Και έτσι έπρεπε να μεριμνήσουμε για σχολεία. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζουμε εδώ και 7 χρόνια ως ε, ε, μητροπολιτική ζώνη του Γκαζιαντέπ. Ανοίξαμε μάλιστα και ένα κέντρο ε, το οποίο για να το ανοίξουμε κάναμε την έρευνα. Τι χρειάζεται, τι χρειάζεται μια κοινωνία ή μια κοινωνική ομάδα για να μπορέσει να ενταχθεί στην κοινωνία υποδοχής. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια πιο αρμονική συμβίωση. Κάναμε λοιπόν την έρευνα πρώτα για να ανοίξουμε το κέντρο αυτό που εξυπηρετεί τις κοινωνικές πολιτικές. Με μια σειρά από μαθήματα που προσφέρουμε σε γυναίκες, πρόσφυγες, σε παιδιά, για να αποτρέψουμε την κετοποίηση, Η η οποία οπωσδήποτε έχει σαν επόμενο βήμα την ε, ρίζοσπαστικοποίηση αυτό ήταν ο γνώμονας με τον οποίο προχωρήσαμε. Προσφέραμε μαθήματα γλώσσας, προσφέραμε μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης και πάνω απ' όλα θελήσαμε να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανθρωπιά την δυνατότητα να αναπτύξουν το δυναμικό τους. Και βεβαίως Πρώτος στόχος μας ήταν να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τα παιδιά, γιατί έχουμε αυτήν την θεμελιώδη ε, φιλοσοφική προσέγγιση που άλλωστε είναι κοινή με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η γυναίκα, το παιδί πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη φροντίδα και περιποίηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε με την υποστήριξη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προχωρήσουμε σε ταχύτερη εξασφάλιση των αναγκών ε, και της υποστήριξης που χρειάζεται, μέχρι και παιδικού σταθμού, σε την μπορέσαμε να ανοίξουμε και διατηρούμε. Το Gaziantep, ε, για να σας δώσω μια εικόνα ε, σε αδρές γραμμές, υποδέχτηκε μέσα στην τελευταία επταετία πληθυσμό μεταναστών και προσφύγων ισοδύναμο με αυτό, τον Βρυξελ, το, με το, με αυτό του 50% του πληθυσμού των Βρυξελών. Καταλαβαίνετε τι σήμαινε αυτό και σε όρους ε, παρεχόμενης στέγης και λοιπόν υποδομούν 17.000 μόνο είναι τα παιδιά τα οποία είναι ε, ανήλικα και υποδεχόμαστε κάτω από 18 ετών δηλαδή. Με σχολεία τα οποία έχουμε προσφέρει εμείς, τα οποία έχουμε οργανώσει ε, κατά τρόπον ώστε το 67% τουλάχιστον των παιδιών ε, μπόρεσαν να ε, μπουν στο σχολείο μέσα στην πρώτη τετραετία από την, άφηξη, από την εκκίνηση του φαινομένου αυτού. Πρέπει να σας πω ότι τα ποσοστά τα οποία έχουμε επιτύχει, τα ποσοστά προσφοράς παιδείας και εκπαίδευση στα παιδιά αυτά είναι ισοδύναμα με αυτά που θα είχαν, αν όχι καλύτερα, με αυτά που θα είχαν στην στην πατρίδα. Αν είχαν μείνει στη Συρία δηλαδή, θα είχαν τα ίδια ποσοστά ε, ε, παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο. Το ίδιο σε σχέση και με την εργασία και απασχόληση. Έχουμε ξεκινήσει ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει την εξασφάλιση θέσεως εργασίας χωρίς ποσοστώσεις, χωρίς αποκλεισμούς στους υποψηφίους εργαζομένους. Και έτσι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ σημαντικό ε, πρόγραμμα. Έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο πρόγραμμα επίσης με ε, κανάλια αρδευτικά, 120 χιλιόμετρα συνολικά, ε, το οποίο εξασφαλίζει την ίδρευση, την άρδευση και γι' αυτό το λόγο σας λέω ότι μιλούμε για ένα συνολικό μοντέλο του Γκαζιάντεπ. Είδατε πόσο πυλισχυδές είναι αυτό. Ουσιαστικά χρειάστηκε να χτίσουμε μια καινούργια πόλη. Γιατί, Γιατί έφτανε πολύ ε, υψηλά το ενίκιο στα υφιστάμενα, στην υφιστάμενη στέγη, καθώς υπάρχει και ε, παρουσία στρατιωτική στην περιοχή και άρα ε, αυτό ούτως ή άλλως ε, πίεζε προς τα πάνω τα ενίκια. Χρειάστηκε λοιπόν να φτιάξουμε καινούρια στέγη, να χτίσουμε καινούριε κατοικίε. Εμείς για να σας εξηγήσω την προσέγγιση μα, την μετανάστευση την είδαμε σαν ένα αποτέλεσμα, όχι σαν ένα αίτιο. Ότι δηλαδή, αν υπάρχουν αυτέ και αυτές οι συνθήκες τότε υπάρχει πίεση μεταναστευτική. για οποιονδήποτε μπορεί να διαμαρτύρεται για τη μετανάστευση, θα συνιστούσα να κοιτάξει ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους κάποιος άνθρωπος αφήνει το σπίτι του και μεταναστεύει. Κοιτάξτε τη Μέση Ανατολή όχι ως μια πηγή πετρελαϊκών πόρων, όχι ως ένα διάβλο των μεγάλων αγωγών του πετρελαίου. Κοιτάξτε την σαν μια πηγή ε, ανθρώπων ε, με δυνατότητες που έχουν ανάγκη από ενσωμάτωση στις κοινωνίες που μπορούν να αποτελέσουν το για όλες τις κοινωνίες όπως αποδείχθηκε και για τον Τεπ. Η συζήτηση ε, που κάνουμε σήμερα ε, είναι πολύ σημαντική και γιατί μας επιτρέπει να ε, μιλήσουμε για τον Gaziantep, για τα προγράμματα, τα εθελοντικά που αναπτύχθηκαν, αλλά ταυτόχρονα τονίσουμε και το γεγονός ότι η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζωτική σημασία για μας γιατί εξασφαλίζει μια σταθερότητα στις ροές Οπωσδήποτε είναι πολύ σημαντικό αυτό που ακούστηκε νωρίτερα ότι πρέπει να ε, δοθούν δυνατότητες για νόμισμη μετανάστευση. Πρέπει η μετανάστευση όμως να δώσει δυνατότητες όχι μόνο σε αυτόν που είναι εποφελής ή χρήσιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δώσει δυνατότητες και, στον, ε, και στο παιδί, το ορφανό, τον ηλικιωμένο, τον άρρωστο. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να χαθεί ανθρωπιά από τον κόσμο. Αυτή είναι η δική μου η έκκληση. Ε, η δική μου έκκληση, σας μιλώ ως γυναίκα, σας μιλώ ως άνθρωπος, να ανοίξουμε τις αγκαλιές μας, να δείξουμε μια πιο ανθρώπινη, ε, ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει την αγκαλιά της και να υποδεχθεί περισσότερους ανθρώπους. Αυτά ήθελα να σας πω για το μοντέλο του Γκαζιαντέπ, να μοιραστώ μαζί σας και κυρίω να μιλήσω για την ανθρωπιά, για το δίκαιο του ορφανού, για το δίκαιο της γυναίκας, για το δίκαιο του ηλικιωμένου. Και ελπίζω, ελπίζω και πιστεύω ότι πρέπει να αναλυφθούν αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε κάθε περιοχή του κόσμου. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε κυρία Δήμαρχε Σαχίν. Σας ευχαριστούμε που μας παρουσιάσετε την εμπειρία τη δική σας και της περιοχής σας. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε και τις ε, εμπειρίες άλλων εθνικών βουλευτών που ήρθαν εδώ για να τις μοιραστούν μαζί μας. Σας ευχαριστούμε θερμά πάντως για τις παρουσιάσεις σας μέχρι τώρα. Εκτιμούμε ιδιαίτερα σε όλη αυτή την προσπάθεια. Τώρα απευθύνομαι στην Ομίγυρη. Ευχαριστώ καταρχήν για την εμπιστοσύνη ομιλητών. Η κυρία Ντάναη από το ΕΛΚ της Ουγγαρίας είναι η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Μόνικα Ντανάη από το ΕΛΚ και την Ουγγαρία. Παρακαλώ δύο λεπτά έχετε στη διάθεση. Αξιότιμοι συνάδελφοι εκ μέρους της ε, Ουγγρικής κυβέρνησης, ε, θα ήθελα να σας πω τα εξής. Ότι η Ουγγαρία έχει να δώσει διαφορετικές άλλες απαντήσεις από αυτές που δίνουν κάποια. Ό,τι αφορά τους πρόσφυγες έχουμε νομικές υποχρεώσεις, όσον αφορά τους μετανάστες εκεί ισχύει κάτι άλλο και ευχαριστώ τον εισηγητή των Μερών Εθνών που όσον αφορά τα Γκαζιαντέπ και έχω πάει εκεί. Θέλω να συγχαρώ ε, την κυρία Δήμαρχο για το εξαιρετικό της έργο. Έχουμε να κάνουμε πιο πολύ υπάρξει ένας ε, μηχανισμός ώστε να γίνει ανακατανομή του βάρους ε, όσον αφορά την μετακατάσταση Και η Ουγγαρία πρέπει όσοι μας με τις συμφωνίες επανεισδοχής και τις συμφωνίες γενικότερα όπως ε, δεν υπάρχει ε, λιβική υπάρχουν αντάρτες και ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό και με αυτές τις συμφωνίες ε, ενισχύουμε την ε, λαθροδιακίνηση. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε και θα ήθελα να ρωτήσω τους συναδέλφους από το Εθνικό Κοινοβούλιο, από χώρες που έχουν το σύστημα, τα προγράμματα των ε, χορηγών επενδυτών, τις χρυσές θεωρήσεις. χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την ε, δημογραφική μείωση στην Ευρώπη, παρά, παράλληλα όμως δίνουν χρυσές θεωρήσεις σε πλούσιους μετανάστες, πολλοί από τους οποίους που θέλουν να σε πλούσιους μετανάστες, πολλοί από τους οποίους που θέλουν να ε, δραστηριότητες. Μάρτιν. Χωσέ Αλβέρτο Μάρτιν Τολεδάνο από την Ισπανία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Γκονσάλες. Δεν θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα που είπε ότι δεν και εσύ προσπαθώντας να γλιτώσουν από τη βία ή από τη δολοφονία. Αυτό είναι τραγωδία και είναι και πρόβλημα. Και πρόβλημα είναι και η διέλευσή τους ε, όταν έχουν βάλει πορεία προς την Ευρώπη το βόρειο ημισφαίριο, γιατί διέρχονται από χώρες ε, που παραβιάζουν τα δικαιώματά τους στις χώρες άφηξης, στις χώρες προορισμού, γιατί οι χώρες μας δεν είναι έτοιμες ούτε από πολιτική νομοθετική, ούτε από κοινωνική άποψη, ούτε και άποψη νοοτροπίας για τόσο σημαντικές μαζικές μερικές φορές ροές ανθρώπων που θέλουν να βελτιώσουν τις βιωτικές τους συνθήκες. Γι' αυτό και στην Ισπανία που ε, νομοθεσία ε, με μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν πρώτες το πρόβλημα και θα πρέπει να αναζητήσουμε αλληλέγγυες λύσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Επίσης, ε, κρίνουμε πολύ σημαντικό την παράλληλη επεξεργασία διαφόρων θεμάτων των ανθρώπων αυτών στις δικές μας κοινωνίες. Εγώ ελπίζω πάντως ότι το έργο και η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει αίσιο αποτέλεσμα, ώστε να έχουμε μια πολύ ε, πιο τυπική, νομότυπη και μετανάστευση που πραγματικά θα... Τα προβλήματά μας έχουν δημιουργηθεί κυρίως ε, από την παράτυπη, παράνομη μετανάστευση από το 2015 που είχε μαζικές διαστάσεις και έδειξε πόσο προετοίμαστε ήταν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν αυτό το φαινόμενο. Δεν θα σχολιάσω τις ε, μεμονωμένες παρατηρήσεις ε, της Γερμανίδας Καγκελαρίου ή τις ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που δεν ήταν πάντοτε οι πιο κατάλληλες και οι πιο σωστές. Πάντως νομίζω ότι ε, συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να αναχαιτήσουμε την άφηξη παράνομων μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προετοιμαστούμε για τις νόμιμες μεταναστευτικές ροές με σωστή διαχείριση βέβαια. Ε, σε ό,τι αφορά τη χορήγηση της ηθαγένειας, ε, τα κράτη-μέλη είναι κυρίαρχα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει Ευρωπαίους πολίτες, δεν έχει Ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Τέτοια ε, αρμοδιότητες υπάρχουν σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη χορηγούν υπηκότητα, ηθαγένεια και τα κράτη φροντίζουν για τους πολίτες τους. Δεν θα πρέπει να επεμβαίνει στη διαδικασία αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να σέβεται το δικαίωμα και την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών που θα μπορούν και θα πρέπει να λαμβάνουν κυρίαρχα τις αποφάσεις τους. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ε, τι ε, αριθμούς μεταναστών μπορούν να απορροφήσουν τα κράτη-μέλη. Και θα ήθελα όλη αυτή η κοινωνική μηχανική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Ηνωμένων Εθνών να μην επιβάλλουν στα κράτη-μέλη ποσοστώσεις ή οράματα που είναι απαράδεκτα για τους λαούς των κρατών μέλων. Θα πρέπει να σεβαστούμε και τη γνώμη της κοινή μας γνώμης. Γιατί ε, αυτούς εκπροσωπούμε στην διαμόρφωση των ανθρώπινων πολιτικών και η γνώμη θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Η κυρία Σπινέλη, παρακαλώ. Σωστές. Και θέλω επίσης να ευχαριστήσω την, Υπουργό, την ε, Δήμαρχο του Γκαζιάντεπ για την ιδιαίτερη προσπάθεια, για... ιδιαίτερα προς τη Δήμαρχο του Γκαζιάντεπ. Θα απευθύνω μια ερώτηση σε μεγάλα ποσοστά αξιοποίηση εργασίας ανηλίκων και παιδιών στην κλωστοϊφαντουργία, ίσως όχι ακριβώς σε παράνομη εργασία απασχόλησης, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα φαινόμενο που έχει πάρει διαστάσεις Ευχαριστώ. Τρία χρόνια μετά το... Το μικρόφωνο σας αν θέλετε στρίψτε το προς σας. Ευχαριστώ πολύ. Το 2015 μπορούμε να συζητάμε αλλά όχι να επαναπαυόμαστε πρέπει να συζητήσουμε για μια βασική αντίφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την αναγνώριση του δημογραφικού προβλήματος και τη του πληθυσμού της Ευρώπης και κατ' επέκταση του εργατικού δυναμικού, την προσπάθεια χρηματοδότηση της ένταξης προσφύγων και μεταναστών και από την άλλη την ενίσχυση της φύλαξη με πρόσχημα την ασφάλεια αλλά και την άρνηση πολλών χωρών στην υποδοχή προσφύγων και μεταναστών και μάλιστα ε, χωρών που έχουν μεγάλο αριθμό μεταναστών σε άλλες χώρες. Θα συμφωνήσουμε με την προσέξη του κυρίου Μοράλες και τις ανησυχίες του. Όντως υφίστανται τα προβλήματα αυτά και το λέω ως μόνιμος κάτοικος ε, της Λέσβου και ενεργό μέλος του τοπικού κινήματος για την υποδοχή προσφύγων και μεταναστών εδώ και πάρα πολλά χρόνια διότι η μετανάστευση στην περιοχή μου υφίσταται εδώ και δεκαετίες. Η υποδοχή και η υπεράσπιση των προσφύγων που καταφθάνουν εδώ και πολλά χρόνια στη Λέσβο λοιπόν ε, είναι ο δρόμος ε, που παρουσίασε η Δήμαρχος του Γκαζιέντε. Το κάνουμε και εμείς στον τόπο μας αυτό. Αυτός είναι ο ορθός δρόμος και με τρομάζει η άρνηση πολλών ε, συναδέλφων να ακούσουν αυτόν τον δρόμο. Αρνούνται να ακούσουν. Να πάνε και να δούνε τι γίνεται και να έρθουν και στη Λέσβο να δούνε κομμάτια της ένταξη στα σχολεία, ε, στις δημόσιες, ε, την, πρόοδο στη δημόσια υγεία που βοήθησε και τον τόπιο πληθυσμό τελικά η ενίσχυση αυτή. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ε, με ένα παράδειγμα της κόρη μου που σήμερα είναι 6 αλλά το καλοκαίρι του 15 ήταν 3,5 στην ερώτησή της τι γίνεται με τους ανθρώπους που έρχονται από τη θάλασσα και γιατί έρχονται από τη θάλασσα και στην απάντησή μου ότι γίνεται πόλεμο στον τόπο και αναγκάζονται να φύγουν, η αθότητα ενός παιδιού είπε ότι πώς κάνετε έτσι. Να φτιάξουμε μια πιο μεγάλη και πιο γερή μυτιλίνη να χωρέσουμε όλοι. Αν εμείς ως ενήλικοι το μεταφέρουμε αυτό στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο δρόμος που μπορούμε να βρούμε για μια σύγχρονη Ευρώπη. Για τις τη θα πρέπει να επεκταθεί και στα αδέρφια. Αυτό κατά την άποψή μα είναι αντιπαραγωγικό, όπω και η δυνατότητα. Θα πρέπει επίση τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ασφαλή και αυτό το υποστηρίζουμε και επίσης το γεγονό ότι υπάρχει το σχέδιο για ε, ζώνες με ε, αφορά την ε, χορήγηση στάτους ε, πρόσφυγα. Ευχαριστώ πολύ. του ασύλου όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Έχουμε μακροχρόνια εμπειρία Έχουμε 350.000 ε, ξένους ανθρώπους που εργάζονται στην ε, περιοχή μας ως ερευνητές, ε, έχουμε φοιτητές και πολλούς από αυτούς με τα κρατημέλη. Αυτά θα αποφασίσουν ποιος θα προσκληθεί στην αγορά εργασία τώρα όσον αφορά... Τα 60 εκατομμύρια ανθρώπων Ε, στα σημεία στα οποία ήδη βρίσκονται. Κάνουμε λόγο για την κατάσταση στις πιο ευάλωτες ομάδες ανθρώπων, όπως είναι τα παιδιά, ε, σε κέντρα που δεν έχουν την σωστή ιατρική φροντίδα. Το 2015 η κατάσταση είχαν αρκετά χρήματα και δύναμη για να μπορέσουν να το πράξουν αυτό και τους πιο ευάλωτους, όπως είναι οι γυναίκες και τα παιδιά, Του αφήσαμε εκεί που ήταν, δεν του δεχτήκαμε. Επομένω η λύση δεν είναι η μετεγκατάσταση, αλλά η Αφρική για την επεξική βοήθεια και τι επενδύσει. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το άνοιγμα τη αγορά με αυτέ τι χώρε. Γιατί η δικιά μας πολιτική ε, ενισχύει την φτώχεια σε αυτές τις χώρες, καθώς οι αγορές μας είναι κλειστές Εκεί κάνουμε λόγο για εξτομικευμένη αξιολόγηση, αλλά όχι για την ε, μαζική μετανάστευση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάνν Σκόπεκ από την Τσεχία στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι πρέπει να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στην παράτυπη μετανάστευση και την ε, ελκυστικότητα που πρέπει να έχουμε, ε, να δείξουμε στους ε, εξειδικευμένους εργαζόμενους. Είναι λάθος να τα συγχαίρουμε αυτά τα δύο, γιατί δεν θα βρούμε μια λειτουργική λύση. Η Τσεχία θέλει να εστιάσει στις αιτίε της μετανάστευσης και όχι μόνο τις συνέπειες και γι' αυτό το λόγο η πολιτική επανεισδοχή θα πρέπει να είναι πιο αποδοτική και να καταπολεμήσει την λαθρεία διακίνηση. Όσον αφορά το σύστημα ασύλου θα πρέπει να ε, βασίζεται στην συνένεση γιατί είναι βάλουμε κανόνες, αυτό μόνο θα εμβαθύνει την κρίση. Ένα ψήφισμα του δικού μας κοινοβουλίου υιοθετήθηκε πρόσφατα και αρνείται ε, την διόρθωση που έχει γίνει στους μηχανισμούς ε, επανεγκατάσταση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να είναι υπεύθυνα για αυτές τις αποφάσεις και θα προσπαθήσουμε να ε, διασφαλίσουμε ότι αν υπάρξουν αλλαγές στην πολιτική ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποστηρίξουμε, θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε την αρχή της ομοφωνίας ώστε το σύστημα ασύλου να μην είναι καταχρηστικά. Ακούγοντας ε, τις ομιλίες σας, κατανόησα ότι η παράτυπη μετανάστευση θα μετατραπεί σε νόμιμη μετανάστευση με απλά διοικητικά μέτρα. Αυτός δεν είναι ο τρόπος να διαχειριστούμε την κατάσταση και για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της γύρασης του πληθυσμού με τη μετανάστευση από άλλες κουλτούρες. Ε, δεν θεωρώ ότι αυτό το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό όσο το παρουσιάζεται γιατί όταν κοιτάζω τα ποσοστά ε, ανεργίας ε, των νέων ε, στις, στα παλιά κρατημέλη δεν θεωρώ ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα. Αγαπητοί συνάδελφοι, έτσι ολοκληρώνεται ο κατάλογος των εκπρόσωπων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ ιδιαίτερως τους προσκεκλημένους μας από τα Εθνικά Κοινοβούλια για τις τοποθετήσεις τους και τη συνεισφορά τους στη συζήτηση. Πρόκειται βέβαια για ένα ζήτημα άκρος ε, δυσχερές και ευαίσθητο. Στο θέμα της, με, της ενσωμάτωσης, επιτρέψτε μου να σημειώσω ότι δεν υπάρχει δυνατότητα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, κοινοβούλιο, επιτροπή να προωθήσουν ενσωμάτωση ένταξης της κοινωνίας. Είναι κατεξοχήν ζήτημα όπου τα κράτη-μέλη, οι περιφέρειες, οι τοπικές αρχές πρέπει να αναπτύξουν τη σχετική δραστηριότητα. Για δε τις νόμιμες οδούς δεν υπάρχουν προτάσεις συγκεκριμένες, το ανέφεραν αρκετοί, είναι λίγες οι προτάσεις, είναι σε δυσκολία ε, και βεβαίως υπάρχουν ε, και οι περιορισμοί του πόσο εφάνταστος και δημιουργικός μπορεί να κάνει στο σχεδιασμό τέτοιων λύσεων και από πλευρά των θεσμικών οργάνων σημειώνω πάλι είναι περιορισμένε οι δυνατότητες. Σας ευχαριστώ λοιπόν θερμά για τα σχόλιά σα και για το ενδιαφέρον ε, για συμμετοχή στη συζήτηση και ευχαριστώ και του ευρωβουλευτέ, βέβαια, ακούσαμε κάποιε φωνέ από του ευρωβουλευτέ μα σήμερα. Ιδιαίτερος, ωστόσο ευχαριστώ του προσκεκλημένου μα τον κύριο Κονσάλε Μοράλε, του εκπροσώπου τη Βουλγαρική Προεδρία. Θα είναι σκληρή και σημαντική οι έξι μήνες της προεδρία σας. Σας ευχόμαι κάθε επιτυχία. Ξέρω ότι έχετε κάνει τεράστια προετοιμασία για αυτό το εξάμεινο. Σας ευχαριστώ πολύ καλοί συνάδελφοι και εύχομαι ό,τι καλύτερο για του επόμενου έξι μήνες, για τους επόμενους έξι μήνες και για την ε, κυρία Μαρχό. Την ευχαριστώ θερμά για όλη τη δουλειά της, για το καλό παράδειγμα που έδωσε, παράδειγμα και ενσωμάτωσης και αποδοχής που μας παρουσίασε σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ και σημειώνω ότι είναι απολύτως αδύνατο να γίνει εις βάθος εξαντλητική, πλήρης και αναλυτική συζήτηση ε, των θεμάτων αυτών στο διάστημα που έχουμε στα θέση μας, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι μπορέσαμε εθνικοί βουλευτές, ευρωβουλευτές, ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα αυτό και άλλοι εκπρόσωποι αρχών να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε. Παρακαλώ τους προσκεκλημένους μας ή δυνατόν να μείνουν, ε, εφόσον τους το επιτρέπουν υποχρεώσεις τους και για το επόμενο κομμάτι της ε, συζήτησης. Από ό,τι μαθαίνω δυστυχώς για το επόμενο κομμάτι η κυρία Νετφέλτ που, θα, που είναι η συγγήτρια και έπρεπε να προεδρεύσει δεν... Α, όχι, με συγχωρείτε. Είχατε κάτι να απαντήσετε νομίζω, έτσι μια ερώτηση. Παρακαλώ. Βεβαίω αν ε, θέλετε να δώσετε σύντομα μια απάντηση. Αγαπητή κυρία Βουλευτά, για το θέμα της εργασίας των παιδιών στην κλωστή φαντουργία που ρωτήσατε, θέλω να επισημάνω το εξής και το είπα και κατά την ομιλία μου, ε, εκεί όπου υπάρχουν ε, ε, μεταναστευτικές ή προσφυγικές ροές, αν δεν αναλυφθούν τα κατάλληλα αποτρεπτικά μέτρα, προφανώς θα καταλήξουν τα παιδιά στην παράνομη εργασία. Εμείς αυτό που προσφέρουμε στα παιδιά και έχουμε καταφέρει να δώσουμε είναι στα, μέχρι τα 16 τους να τα κρατάμε στην εκπαίδευση, να τους προσφέρουμε εκπαίδευση και 70% των παιδιών αυτών που έχουν έρθει ως μετανάστες ή πρόσφυγες είναι σε σχολεία στην Τουρκία μέχρι τα 16 τους. Αν δεν υπήρχε αυτή η πολιτική της Τουρκίας, όχι, θα, όχι θα δουλεύανε παράνομα στην κλωστή τα παιδιά αυτά, θα είχαν μπορέσει να επιζήσουν. Χρειαζόμαστε 6.000 τάξεις σχολικές για να δώσουμε ε, την απαιτούμενη ε, μόρφωση στα παιδιά, στο σύνολό τους, έτσι ώστε να καλύψουμε 100% των παιδιών. Και πρέπει να σας πω ότι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ και αυτό που είπατε για την κλωστοϊφαντουργία. Το παρακολουθούμε και μέσω του Υπουργείου εργασίας και προσπαθούμε και τα παιδιά αυτά να προστατέψουμε και να ενισχύσουμε, να τους προσφέρουμε ό,τι χρειάζονται και βεβαίως να αποτρέψουμε οτιδήποτε κακό και πάντα βεβαίως συμφωνούμε με αυτά που είπατε και σας υποστηρίζουμε. Σας ευχαριστώ. Ε, σίγουρα οι ομιλητές ε, έθεσαν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων. Ε, αν θέλετε συγκεκριμένα ζητήματα να θέσετε προς τους καλεσμένους μας, μπορείτε να στείλετε και γραπτός ε, τα, τις ερωτήσεις και θα λάβετε γραπτός απαντήσεις από τους καλεσμένους. Η κυρία Ιντβελτ που κανονικά έπρεπε να παιδεύσει το δεύτερο σκέλος, ε, γιατί είναι η συγγήτρια για τις συνθήκες ε, της υποδοχής, τελευταία στιγμή ακύρωσε την παρουσία της, οπότε θα χρειαστεί να με υποστείτε για λίγα λεπτά ακόμη. Λυπάμαι, συνήθως γίνεται αλλαγή. Θα προεδρεύσω για λίγα λεπτά ακόμη με τη βοήθεια της κυρίας Κίνγκα Γκάλ, που είναι αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών. Και την ευχαριστώ πάντα για την αμύωτη στήριξή της και στην Επιτροπή και εδώ. Περνάμε στο επόμενο τμήμα της ε, διακοινοβουλευτικής διάσκεψης. Παρακαλώ τους καλεσμένους του επόμενου πάνελ να λάβουν θέση στο Προεδρείο και να σας ευχαριστήσω όλους για την υπομονή σας. Με το που θα συσταθεί το πάνελ θα ξεκινήσουμε τις εισαγωγές και ευχαριστώ και πάλι για την υπομονή που δείχνετε. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ, καθίστε για να συνεχίσουμε. Ξέρω ότι μερικοί έχουν ανάγκη ένα διάλειμμα. Και έξω έχουμε και μηχάνημα διανομής καφέ. Ελπίζω να βοηθά. Και παρακαλώ, επιστρέψτε το Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ θα ξεκινήσουμε το δεύτερο τμήμα της διακοινοβουλευτικής αυτής σύσκεψης. Κάποια στιγμή θα δώσω τη σκητάλη της Προεδρίας στην κυρία Κίνγκα Γκάλ, που είναι αντιπρόεδρος Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, γιατί η κυρία Ιντβελτ που κανονικά έπρεπε να προεδρεύσει, κολλείεται λόγω κάποιας κατεπίγουσας οικογενειακής ε, κατάστασης που προέκυψε. Οπότε θα προεδρεύσω εγώ. Έχουμε το δεύτερο σκέλος, τους νόμους διάβλους για τη διεθνή προστασία. Καλωσορίζω και πάλι για αυτό το τμήμα της ακρόασης ε, του φαινομένου να παίζουν τη ζωή του κορώνα γράμματα χρήζονται σε διεθνή προστασία αναζητώντα κάποιο καταφύγιο. Είδαμε την κατάσταση στη Μεσόγειο, στα νησιά του Αιγαίου, στη Λαμπεντούζα, στην Κεντρική Μεσόγειο, τα, ε, τις διόδους Κεντρικής Μεσογείου. Είδαμε εικόνες ε, ε, για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όλοι παρακολουθούμε αυτά τα θέματα. Είναι τεράστιο το ζήτημα για μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι αντιμετωπίζουμε και το ζήτημα των λαθροδιακινητών και της ε, διακίνησης και καλούμαστε εδώ να βρούμε λύσεις. Βέβαια δεν είμαστε αφελείς, δεν θεωρούμε ότι θα επιλύσουμε σήμερα διαμαγές όλα τα προβλήματα, αλλά αυτή η ανταλλαγή απόψε μεταξύ μας, ε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων έχει κρίσιμη σημασία. Και σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε αυτές τις επαφές μας για αυτό το τόσο κρίσιμο κοινοβούλιο για να να εξετάσουμε ζητήματα όπως η επανεγκατάσταση, η μετεγκατάσταση και άλλα συναφή. Αλλά πολλά από τα θέματα αυτά έχουν γίνει επίμαχα και προβληματικά, δύσκολα, δυσεπίλητα και το θέμα της αλληλεγγύης επίσης. Θα μπορούσα να μακρυγωθεί ότι ε, γίνεται άνευ προηγουμένου έργο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Βουλγαρική Προεδρία πάνω το 40% όλων των νομοθετικών προτάσεων ε, του εξαμήνου αφορούν το ζήτημα αυτό και ένα μεγάλο τμήμα των νομοθετικών τύφωση της νομοθεσίας Γιατί είτε είχαν μείνει ανεφάρμοστε κάποιες νομοθετικές προτάσεις είτε δεν υπήρξε η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί η κρίση, να γίνει σωστή διαχείριση. Και εξού και η σημερινή κατάσταση. Γνωρίζετε και εσείς τα πράγματα και στα Εθνικά Κοινοβούλια. Γνωρίζετε την κρίση που αντιμετωπίζουμε. Τους καλεσμένους μας εμπειρογνώμονες και πρώτα απ' όλα με τιμά ιδιαίτερα που θα δώσω το λόγο στον Πίτερο Σάλιβαν που είναι αρμόδιος για θέματα επανεγκατάστασης στο Γραφείο για την Ευρώπη του, της ΥΠΑ των Ηνωμένων Θα μας κάνει μια εισαγωγή για το θέμα της επανεγκατάστασης και θα ανακατάστασης για το 2018-2019 και μέχρι στιγμής 14.000 έχουν, για 14.000 θέσεις έχουν αναλυθεί δεσμεύσεις, ελπίζουμε να αυξηθούν. Το 2016 ήταν για την ύπατη αρμοστία μια σημαντική χρονιά και είχαμε τη ρεκόρ, χώρισαν ε, για επανεκατάσταση παγκοσμίω. Και ήταν ε, αριθμοί ρεκόρ την τελευταία 20 ετία τα νούμερα αυτά. Το 2016 επίσης είχαμε και τη διακήρυξη της Νέα Υόρκη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ορόσημο ήταν αυτή η διακήρυξη γιατί 193 χώρε του φυγικού και του μεταναστευτικού ζητήματος στο μέλλον. Δυστυχώ και παρά την εφορία που επικράτησε στην αρχή, αυτός ο ενθουσιασμό δεν επικράτησε και τώρα σημαντική μείωση δηλαδή των διαθέσιμων θέσεων επανεγκατάστασης και έτσι ε, υπολοιπόμεθα ε, σε σχέση με τις ανάγκες μας. Θέλουμε περισσότερε είπα. Και θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητε για το 2018. Για παράδειγμα, η προτεραιότητα είναι η Κεντρική Μεσόγειος. Ήδη έχει ε, ασφαλώ στην Ευρώπη. Η πατερμοσία, η αρμοστία ζήτησε 45 επιπλέον χιλιάδες θέσεις. σε, γνωρίζετε, δεδομένης ε, δεδομένων των αντίξων ε, συνθήκων ε, και της πολύ δύσκολη κατάστασης της, και της άμεσης που γίνονται από τη Λιβύη προς την Ιταλία. 162 εκενώθηκαν πέρυσι το Δεκέμβριο. Βέβαια, μέχρι τις αρχές του έτους φέτος και ελπίζουμε να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Σήμερα έχουμε, ε, ζητούμε 40.000 θέσεις σμεύσεις για να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν και στη Λιβύη. Σε ό,τι αφορά τη διακήρυξη της Νέας Υόρκης και το παρά, παράρτημα της διακήρυξης περιλαμβάνει ένα η δέσμευσή μας με τις χώρες αυτές στηρίζεται στον επιμερισμό των ευθυνών και τη διεθνή συνεργασία και σίγουρα η επανεγκατάσταση είναι κέριο σημείο αυτής της συνεργασίας. Και μόνο έτσι το ποσοστό είναι ΣΥΡΙ. Ε, αντιλαμβάνομαι ότι χρησιμοποιώ πολλά στατιστικά στοιχεία που δεν είναι τόσο εύληπτα, αλλά πισμό. αλλά οι ανάγκες όπως σας είπα είναι τεράστιες. Ε, και πολλές άλλες ομάδες πλήν των προσφύγων χρειάζονται επανεγκατάσταση, όχι σύρων ή προσφύγων. Επιπλέον θα ήταν ε, ευχή έργων. Όπως είπα, μέλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη που συνέβαλαν πολύ θετικά σε αυτό το σύμφωνο και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η θετική συνεισφορά. Την τελευταία διετία βλέπουμε για την κινητικότητα των φοιτητών. Θέλουμε να είμαστε καινοτόμοι, ευρηματικοί, ελαστικοί και να ανταποκριθούμε στις τεράστιε ανάγκες που υπάρχουν. Είχαμε σημαντήσει τι ευκαιρίε επανεγκατάσταση, γι' αυτό και ζητούμε τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν αμέριστη την προσπάθειά του στήριξη τη επατησαρμοστία και να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων. Πίτερ, να σα πω πώ θα συνεχίσουμε από εδώ και στο εξή. Θα έχουμε ένα σύντομο βίντεο από την επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Μωρίνο Λάξ, η οποία θα μας μιλήσει για την νομοθεσία ασύλου και πώς εφαρμόζεται. Θα έχουμε εμπειρογνώμονες από εθνικά κοινοβούλια για το Διεθνέ Καθεστώ Προστασία, ε, την κυρία Μαριέτα Καραμαλή από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση, τον κύριο Παρασκευόπουλο από την Ελληνική Βουλή και τον κύριο Μπουστήλ από το Κοινοβούλια της Μάλτας. Τους καλωσορίζω όλους και Θα ξεκινήσουμε με την κυρία μωρένο η οποία είναι επικούρ καθηγήτρια στο Πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου. Στη συνέχεια η Κίνγκα Κάλ θα πάρει την προεδρία. Στη θέση της κυρίας Ιντεβέλ που είχε κάποια οικογενειακά προβλήματα και δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Σε ευχαριστώ Κίνγκα που με βοηθάς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με ένα βίντεο από την ε, καθηγήτρια Μόρενο Λάξ. Ευχαριστώ πολύ και... ...to address the role of pieces for legal avenues. I'd like to do this in five... Για το βίντεο αυτό δεν προβλέπετε διερμηνία. ...on humanitarian visas at EU level are not new. The measure was first thoroughly examined in a study for the European Commission back in 2002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 θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Μαρία. Και πολύ σύντομα. Καταρχάς εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονό ότι η Επιτροπή σας μας επιτρέπει να συζητήσουμε κάποιες πτυχές της μεταναστευτικής πολιτικής που έχουν ε, παραγνωριστεί λόγω της σπευσμένη διαχείρισης μιας κρίσης που ήταν η μεταναστευτική κρίση, αλλά πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα επίγουσα ε, κρίση, αλλά και να εξασφαλίσουμε του όρους εκείνους προστασίας ε, και οργάνωσης από τις μεταναστευτικές ροές που χρειάζονται εξελίξεις στη Λιβύη μας δείχνουν ότι η διάκριση μεταξύ οικονομικών μεταναστών και προσφύγων που θα δικαιούνται ε, άσυλο δεν είναι πλέον ευχερής. Και έχουμε να κάνουμε με συνθήκες όλο και πιο τραγικές τελευταία που δεν μπορούν να περιγραφούν ούτε ως καθαρή οικονομική μετανάστευση ούτε ως αναζήτηση ασύλου. ασφαλής χώρες. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς η μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς ε, προκύπτει στον ε, τομέα της μεικτής αρμοδιότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών μπορεί να οργανωθεί κατά τρόπο ε, κοινό ε, με ενίσχυση βεβαίω και των αρμοδιοτήτων νόμης μετανάστευσης εν τέλει είναι πολύ περιορισμένες είναι πολύ περιορισμένο το φάσμα των απαντήσεων και των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα κράτη-μέλη εν, ώψη του φάσματος των προβλημάτων και των δυνατοτήτων και αναγκών των ανθρώπων αυτών, ανδρών και γυναικών που μπορεί να συμβάλλουν από σημαντικέ πιέσεις. Ε, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι μπορεί κανείς να διατυπώσει και διαφοροποιημένες κρίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές αφήξεις μεταναστών το 2015-2016, αυτά τα κέντρα πρώτης υποδοχής που βεβαίως επέτρεψαν και την καταγραφή ε, που πρέπει να αναπτυχθούν δύο συγκεκριμένα που θα μπορούσαν να αποτρέψουν ε, τον υποψήφιο από την ε, αναχώρηση για αυτό το ε, που αποφασίστηκαν το 2015 σε επίπεδο Συμβουλίου μόνο 80% έχει υλοποιηθεί αλλά πρέπει να ενισχυθεί αυτή η προσέγγιση όπως άλλωστε ζήτησε τον προσφέρονται στην πραγματικότητα και πράξη. Ε, επίσης πρέπει να εξασφαλιστεί ένα σταθερό και εξελικτικό μεταλλασσόμενο στάδιο για τη διευκόλυνση αυτής της εγκατάστασης με εθνούς προστασίας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Είναι κομμάτι του πακέτου ασύλου που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή. Επομένως και επανεγκατάσταση οι λύσεις έδωσε τη δυνατότητα για λύσεις συντονισμένες, για κάποιες λύσεις συντονισμένες. Έτσι λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε, να σχεδιάσουμε έναν ε, μηχανισμό ε, υποδοχής γύρανσης. Χρειάζονται ακόμη περισσότερη οικονομική μετανάστευση. Και του πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να οργανώσει αυτή τη μετανάστευση για λόγους αναζήτησης θέσεων εργασίας αναθευτικών μοντέλων. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να προτείνει ένα κοινό πλαίσιο για συγκεκριμένε μορφές οικονομικής μετανάστευσης που θα διευκολύνει την κινητικότητα των επαγγελματικών δεξιοτήτων τη ε, οικονομικής ανάπτυξη ανάπτυξη στι χώρες προελεύσεω στην ενίσχυση του οικονομικού του δυναμικού. Είναι ιστορικό γεγονός και επαναλαμβάνεται μόνο η αναδιανομή όρους που θα σημάνει οπωσδήποτε ε, και μετριότερες μεταναστευτικέ πιέσεις από τα γειτονικά κράτη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Το άκουσμα των ε, ομιλητών μέχρι τώρα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχουμε μια γενική συμφωνία για τους στόχους και μια διαφορά αλλά όλες οι χώρες συμφωνούν για την ανάγκη να βρεθεί μια χρυσή τομή και να υπάρχει και μια διεθνής συνεννόηση σε αυτό το πεδίο. Στον ευρύτερο χρονικό ορίζοντα, ένας σταθερός ρυθμός μετακινήσεων, γεγονός το οποίο καταρρύπτει τον ισχυρισμό τους πληθυσμούς που αντικειμενικά δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους και να τους δεχτεί με όρους ένταξης και όχι Βεβαίως ε, σε ό,τι αφορά την ε, μετακατάσταση, ο μηχανισμός μετακατάστασης, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός ανακατανομής των προσφύγων κράση, διοικητική κράτηση, καθώς δεν δικαιολογείται κατά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η στέρηση της ελευθερίας για σημαντικό την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Το γεγονός είναι ότι εμφανίζεται μια σημαντική απόκληση με τα μερίδιό τους σε ό,τι αφορά την κατανομή του τους αναλογή να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μετεγκατάσταση όλων των επιλέξιμων υποψηφίων της Αφρικής. Νομίζω ότι η αναθεώρηση του κανονισμού του Δουβλίνου να αποτελέσει αυτή η μεταρρύθμιση σημαντικό κίνητρο ώστε να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές και να μην εναποθέτουν την τύχη τους στα, της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Σε ό,τι αφορά <clears throat> τις ελληνικές ενταξιακές προσπάθειες, αυτό που θα ήθελα να πω των ετούντων άσυλο, είτε περιορισμένοι, που αφορά εκείνου που δεν έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου ή μετανάστες που έχουν εκπέσει από την ομιδομένου, ότι υπάρχει δυνατότητα για τα προσφυγόπουλα να εγγράφονται σε κανονικό σχολικό πρόγραμμα ή να παρακολουθούν και προσωρινες δομέ, δομές γιατί δυστυχώς υπάρχουν μέχρι σήμερα κράτη-μέλη που συνεχίζουν να έχουν κάποιες επιφυλάξει για τους τρόπους με τους οποίους αυτό μπορεί να επιτευχθεί. Κάθε κοινή πολιτική όμως εκ των πραγμάτων αν ακόμη και αν επιζητεί συμβιβασμού μεταξύ των εθνικών πρακτικών συνιστά ταυτόχρονα και έμπρακτη μορφή της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.